Colleagues, let's start. Скъпи колеги, на 8 октомври 2019 година Καλημέρα. Τον Οκτώβριο οι συντονιστές αποφάσισαν να εκδώσουν ε, κάποιες νομοδοτήσεις για την απαλλαγή του προπολογισμού του 2018 των διαφόρων υπηρεσιών, διαφόρων υπηρεσιών του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προθεσμία γνωμοδότηση Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών έχει καθοριστεί 23 Ιανουαρίου. Οι συντονιστές της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών αποφάσισαν στις 8 Οκτωβρίου και τον έκρινε αυτό η Επιτροπή, 21 Οκτωβρίου, να εργαστούν μόνο στην Αγγλική για αυτή τη διαδικασία. Και τώρα θα συζητήσουμε την έκθεση Ματσόλα. Μετά θα ανταλλάξουμε απόψεις με τους σκιώδεις ηγητές και άλλους ευρωβουλευτές που θα επιθυμούν ίσως να παρέμβουν. Η κυρία Walsh έχει το λόγο να παρουσιάσει την έκθεση. Δεν μπορεί να είναι παρούσε συνάδελφος ή Τη γνωμοδοτήσεις για την απαλλαγή, συμμετέχει σε αποστολή στη Μάλτα τη ΛΥΜΠΕ. Μου ζήτησε να παρουσιάσω κάποια σημεία. Το σχέδιο γνωμοδοτήσεως παρουσιάζει σήμερα και Ματσόλα παρουσιάζει τι υπηρεσίε Europol, Eurojust, Frontex, Υπηρεσία Θεμελιών Δικαιωμάτων, ΣΕΠΟΛ, ΕΣΑ, ISO και ΟΥΛΙΣΑ και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για τα δεδομένα, προστασία δεδομένων. Σχέδιο γνωμοδότηση έχουμε για την εφαρμογή του προπολογισμού, για την εκτέλεση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτο 2018. Όσον αφορά αυτού του τομεί που εμπίπτουν στην εντολή τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στα πλαίσια τη οριζόντιας, του οριζόντιου σχεδίου γνωμοδοτήσεω για το οικονομικό έτο 2018 εν γέννη, το ελεγκτικό συνέδριο έχει εκδώσει σαφεί γνωμοδοτήσει και για του 10 φορεί που αφορούν αυτή την Επιτροπή, όμως υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν γενικά, κυρίως σχετικά με τη δημοσιο... τις διαδικασίες διαγωνισμών να καταστούν πιο διαφανείς, να μειωθεί εξάρτηση σε εξωτερικά συμβαλόμενα μέρη για πληροφορική, βασικός τομέας αυτός, και να δημοσιεύονται οι κενές θέσεις με τη χρήση της πύλης ε, της ΕΠΣΟ. Η συγγήτρια θέλει να συνεργαστεί με τους και προσβλέπει τι διαπραγματεύσει. Αυτά λοιπόν λέει στο σημείωμά τη η Ρομπέρτα Ματσόλα που πρέπει να είναι στη Μάλτα. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Βόλς. Και τώρα οι σκιώδεις ηγητές έχουν το λόγο και αν το επιτρέπει ο χρόνος στους άλλους ευρωβουλευτές που ίσως θέλουν να πούν κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Ματσόλα για τη δουλειά που έκανε, για τις νομοδοτήσεις. Όπως αναφέρθηκε συνολικά, μόνο μικροπροβλήματα βρήκαμε, αλλά ουσιαστικά στον προϋπολογισμό και στα λογιστικά των υπηρεσιών για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη ε, είχαμε θετική άποψη. Οι απολογισμοί υπήρξαν θετικοί. Εν συντομία, θέλω να αναφερθώ στη δραστηριότητα και για το Eurojust και για την Europol, διότι και οι δύο οργανισμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί οργανισμοί για τα προβλήματα που αφορούν την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια και που αντιμετωπίστηκαν τελευταία χρόνια στο τομείς αυτούς. Είναι σημαντική η κατάσταση Eurojust που πρέπει να συνεργαστεί με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα για καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Σημαντικό και θετικό είναι το έργο και η χρήση των πόρων από το Europol, Europol που εκλήθη να γίνει θεμελιώδης φορέας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας και του κυβερνοεγκλήματος. Σημαντική είχαμε αύξηση των δραστηριοτήτων και αυτό ανταποκρίνεται και σε μια αύξηση σημαντική του προπολογισμού. Λοιπόν, μικροπροβλήματα εντοπίσαμε, όμως δεν βρήκαμε σημαντικά προβλήματα. Τα μικροπροβλήματα μπορούν να διορθωθούν εντάχει να ενθωθώ στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Τοξικομανίας και Ναρκωτικών. Τον περασμένο μήνα, τον Οκτώβριο, πήγα σε αποστολή για λογαριασμό της Επιτροπής πολιτικών ελευθεριών και διαπίστωσα για μία ακόμη φορά και σε αυτή την περίπτωση πως το παρατηρητήριο εφάρμοσε πολύ σοβαρή στρατηγική μέχρι το 2025, έχει επεξεργαστεί στρατηγική με το 2025 με συγκεκριμένους στόχους και έτσι η Ευρώπη θα καταστεί πιο ασφαλής και κατά κάποιο τρόπο πιο υγιής. Διότι ξέρουμε ότι δυστυχώς το θέμα της εξάρτησης από τα ναρκωτικά που γραμμίστηκε από τη διευθύντρια της Europol, Κατερίν Ντεμπόλ, είπε ότι το εμπόριο ναρκωτικών είναι μία από τις βασικές πηγές ε, χρηματοδότησης τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Και έχουμε εκ νέου προβλήματα στον τομέα αυτό, διότι θα θέτει νέες ουσίες στην αγορά, ιδιαίτερα επικίνδυνες μεταξύ άλλων. Τέλος, και κλείνω με αυτό που λέω, για την ΕΑΖΟ. Όσον αφορά την ΕΑΖΟ, δεν μπορούμε να αναφερθούμε στα λογιστικά και στη διαχείριση και να σχολιάσουμε αυτό που είπε το ελεκτικό συνέδριο για το πρόσφατο παρελθόν. Η νέα δίκηση με τη νέα την Ίντα Γκρεγόρη, την νέα εκτελεστική διευθύντρια, δίνει μια αλλαγή και συνεπώς μια προφανή βελτίωση της καταστάσεως και λόγω της νέας διαχείρισης για την εξυγίανση του φορέα και να γίνεται σωστή διαχείριση και διαφανής. Από την πλευρά μου θα πω ότι θα είμαι άκρο συνεργάσιμη. Μέσω τροπολογιών μπορούμε να εμπλουτίσουμε το τελικό κείμενο των γνωμοδοτήσεων συνεργαζόμενοι με τη βασική συγγήτρια την οποία ευχαριστώ εκ νέου για την δουλειά που έκανε. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπρίτσμεντ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ την ε, κυρία Μετσόλα, την εισηγήτρια, για τις 11 γνωμοδοτήσει, το σχέδιο 11 γνωμοδοτήσεων, που θα πρέπει να συζητήσουμε σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να τις διεκπαιρεώσουμε. Είναι πολύ σημαντική διαδικασία απαλλαγής για να ελέγξουμε τον προπολογισμό της Ένωσης και να υπάρχει διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέναντι στους πολίτες. Αυτός ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικός, ειδικά όταν ελέγχουμε τους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνους που εμπίπτουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, θα πρέπει να δούμε το παράδειγμα και να υπάρχουν 100% καθαροί λογαριασμοί ελέγχου. Θα πρέπει να σεβόμαστε τις διαδικασίες. Καλωσορίζουμε τα σχέδια προτάσεων και παρότι που έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, ε, δεν, γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Βασικά το θέμα για μας είναι περισσότερη διαφάνεια για τους οργανισμούς, ειδικά για τη Frontex και τη Europol. Ίσως έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και για τις δύο αυτές νομοδοτήσεις, για την Frontex και τη Europol δηλαδή. Θα πρέπει να κοιτάξουμε με λεπτομέρειες την συνολική γνωμοδότηση που αφορά την ΕΑΖΟ και θα θέλαμε περισσότερες αναφορές στην ΦΡΑ, στην Υπηρεσία Θεμελιδών Δικαιωμάτων, γιατί έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ακριβώς για την επιτήρηση των θεμελιδών δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις και κάποια προβλήματα στη γνωμοδότηση ε, για τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Θέλουμε μια ισορροπημένη γνωμοδότηση και να δείξουμε τις ε, διαδικασίες που έκαναν οι οργανισμοί αυτοί μετά την απαλλαγή του 2017 και το κατά πόσον ακολούθησαν τις συστάσεις. Θέλουμε να βοηθήσουμε το Κοινοβούλιο ε, σε αυτόν τον τομέα, στη δουλειά που κάνει και προσβλέπουμε στην συνέχιση της διαδικασίας. Ευχαριστούμε την κυρία Μπρίτσμεντ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο σκιώδη ηγητή στην αίθουσα. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Κανείς. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 10η Δεκεμβρίου, στο τέλος της εργάσιμης μέρας. Сега ще направим до 9.45 кратко прекъсване и ще продължим с точка. Και τώρα θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι σε 10 παρατέταρτο και θα συνεχίσουμε με το σημείο 20 της μερικής διάταξης. But

So, those of you. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι βρίσκεστε στην αίθουσα, θα σας παρακαλώ να συγκεντρωθούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης. Να εξηγήσω στα μέλη ότι έχουμε εξαιρετικούς τους προσκεκλημένους επιρρογνώμονες Δυστυχώς ε, δεν ε, είναι εδώ όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Θα ήταν ε, χρήσιμο και ωφέλιμο πιστεύω για αυτούς. Βέβαια αυτό οφείλεται στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αποστολή στη Μάλτα και αρκετά μέλη έχουν μεταβεί εκεί. Η αποστολή αυτή εγκρίθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο από το Προεδρείο, γι' αυτό και λείπουν τόσα μέλη σήμερα. Είναι λοιπόν σε μια διερευνητική αποστολή στη Μάλτα αρκετά μέλη της Επιτροπής μας, όμως ας προχωρήσουμε στο σημείο 20 για την τρέχουσα κατάσταση της εφαρμογής του συστήματος εισόδου-εξόδου και του αίτια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότηση Ταξιδιού. Θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά θα γίνει παρουσίαση των εκθέσεων από τον Κρουμ Γκαρκόφ, εκτελεστικό διευθυντή της Ιουλίσα. E Καλώς ήρθατε. Έπειτα θα έχουμε μια παρουσίαση από τον κύριο Ράμο, αναπληρωτή διευθυντή ικανοτήτων της Ευρωπόλ για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης και στο τέλος θα έχουμε ξανά μαζί μας τον Φαμπρίς Λεζερή, εκτελεστικό διευθυντή της Frontex. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξέρετε πως Βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο. Έχουμε να κάνουμε με την εξέταση και τον έλεγχο της ε, εφαρμογής νομοθεσίας και εξετάζουμε λοιπόν το σύστημα εισόδου, εξόδου και το σύστημα πληροφοριών και αδειοδότηση ταξιδιού. Αίτιας είναι πολύ σημαντικά και τα δύο. Γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε αμέσως. Θα δώσω 5-10 λεπτά στον κύριο Γκαρκόφ για την παρουσίασή του και μετά θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι. Πρώτα όμως έχει το λόγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον κύριο Μάρξ Λιόν, επικεφαλής πληροφορικών συστημάτων. Έχετε το λόγο κύριε Σουλών. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή σας που μας έδωσε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για την εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου και του συστήματος αίτιας. Τα δύο αυτά συστήματα εγκρίθηκαν από τους συνομοθέτες αρκετό καιρό πριν με τον κανονισμό για το σύστημα εισόδου-εξόδου που εγκρίθηκε Δεκέμβριο 2017 και τον κανονισμό για το αίτιας που εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ το 2018. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο της εφαρμογής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενεργή στο, στην οργάνωση και ανάπτυξη του συστήματος και οι συνομοθέτες μας ζήτησαν ε, μια σειρά εκτελεστικών πράξεων και πράξεων κατά εξουσιοδότηση για την εφαρμογή του συστήματος. Σε ό,τι αφορά το σύστημα εισόδου-εξόδου υπάρχουν 14 εκτελεστικές πράξεις που αναμένεται να εγκριθούν. Από αυτές 10 είναι ήδη εγκεκριμένες, τώρα που μιλάμε και οι υπόλοιπε είναι αναγκαίε για να τεθεί σε ισχύ εφαρμογή του συστήματο. Οι υπόλοιπε λοιπόν τέσσερι εκτελεστικέ πράξει θα εγκριθούν τους ε, τέσσερι μήνε που μας έρχονται. Δεν είναι απαραίτητη για την ε, λειτουργία του συστήματος, όμως ε, πρέπει να έχουν εγκριθεί πριν. Σε ό,τι αφορά το σύστημα εισόδου-εξόδου, έχουμε επίσης ένα εγχειρίδιο, το οποίο καταρτίζουμε αυτή τη στιγμή για τους χειριστές του συστήματος και για τις αρμόδιες αρχές οι οποίες θα έχουν επίσης πρόσβαση. Επίσης συνεργαζόμαστε στενά με τους αναλυτές για να δούμε τον αντίκτυπο του συστήματος εισόδου-εξόδου στους συνοριακούς ελέγχους. Η θέση σε ισχύ του συστήματος εισόδου-εξόδου προβλέπεται για το πρώτο τέταρτο του 2022. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αίτιας. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εκτελεστικών πράξεων και πράξεων κατά εξουσιοδότηση που εκκρεμεί έγκρισή τους. Έχουμε 13 πράξεις κατά εξουσιοδότηση και 16 εκτελεστικές πράξεις. Είναι αρκετή δουλειά όπως καταλαβαίνετε. Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να αναλύσουμε τη σχέση μεταξύ του αίτιας και των υπόλοιπων συστημάτων, να δούμε δηλαδή πώς μπορεί το αίτιας να ενσωματωθεί στο σύστημα εισόδου-εξόδου και στα υπόλοιπα συστήματα. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε το τεχνικό σκέλος και να φροντίσουμε έτσι ώστε να υπάρχει μία συμμετρία. Σε ό,τι αφορά τις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση, τρεις έχουν εγκριθεί πλήρως. Τρεις είναι σταθερές, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε ήδη μια συμφωνία ως προς το περιεχόμενο, δεν έχουν όμως ακόμα εγκριθεί. Και τέσσερις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, οι οποίες ε, πρόκειται να σταθεροποιηθούν τις ερχόμενες εβδομάδες. Οι τρεις τελευταίες θα εγκριθούν λίγο πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. 16 λοιπόν εκτελεστικές πράξεις μένει να εγκριθούν. 8 από αυτές είναι σταθερές, 3 θα είναι έτοιμες τις ερχόμενες εβδομάδες και οι τελευταίες 5 λίγους μήνες πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. Η έναρξη λειτουργίας του συστήματος αίτιας έχει προγραμματιστεί για τους τελευταίους τρεις μήνες του 2022. Είναι κομμάτι της νέας δομής ενός ε, συστήματος μεγάλης κλίμακας πληροφοριών που θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα αυτά είναι απόλυτα διασυνδεδεμένα, εγγυημένη δηλαδή διασυνδεσιμότητα, και κατά το στάδιο εφαρμογής των συστημάτων αυτών εξετάζουμε την εφαρμογή του κανονισμού διαλειτουργικότητας. Έχουμε δει λοιπόν ότι ορισμένα από αυτά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει προοπτική διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα. Τώρα, η εφαρμογή και των δύο συστημάτων αυτών στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας είναι κάτι το περίπλοκο. Αυτό που, αυτό που απαιτείται από τα κράτη-μέλη είναι αρκετοί πόροι και εργατόρες. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα μηχανισμό ελέγχου της εφαρμογής και των δύο συστημάτων σε επίπεδο οργανισμών, όσες ε, δηλαδή υπηρεσίες και οργανισμοί εμπλέκονται στην ε, κατάρτιση, δημιουργία και λειτουργία του και αναμένεται να είναι έτοιμη την κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη χρήση των συστημάτων αυτών. Να σας υπενθυμίσω ότι και στους δύο κανονισμούς που αφορούν το αίτιας και το σύστημα εισόδου-εξόδου υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις σχετικά με το με την υποχρέωση δήλωσης όλων των κρατών μελών ότι θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν λειτουργία ταυτόχρονα. Αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη-μέλη προχωράνε με τον ίδιο ρυθμό προς την ε, θέση ισχύ του συστήματος σύμφωνα με το προγραμματισμένο, τις προγραμματισμένες ημερομηνίες. Αυτή η παρακολούθηση αποτελείται από τακτικές επισκέψεις στις πρωτεύουσε και σε υψηλό επίπεδο, μεταξύ, άλλος, μεταξύ άλλων. Τα κρατημέλη έχουν κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και ο μηχανισμός παρακολούθησης επίσης θα οδηγήσει σε μία έκθεση η οποία θα περιγράφει την κατάσταση στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μοιραστούν φέλτιστες πρακτικές και τα κράτη-μέλη να εμπνευστούν το ένα από το άλλο για να ολοκληρώσουν τις εργασίες ε, προς την λειτουργία των συστημάτων. Έχουμε ήδη εντοπίσει ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που χρειάζεται να βελτιώσουν την εφαρμογή του συστήματος. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με αυτά και τους έχουμε ζητήσει διορθωτικά μέτρα έτσι ώστε να είναι έτοιμοι στην ώρα τους. Παρακολουθούμε λοιπόν στενά τις εργασίες έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα είναι έτοιμοι ταυτόχρονα. Για να ξεκινήσει η λειτουργία του συστήματος εισόδου-εξόδου που προβλέπεται για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Και η έναρξη λειτουργίας του αίτια στο τελευταίο τρίμηνο του 2022. Σας ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Το κύριο Σκάρτοφ, Γενικός Διευθυντής. Έχετε το λόγο. Καλημέρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθούμε στην πρόοδο που έχουμε κάνει όσον αφορά το ESM και το ETIAS. Το έργο του Ελίσσα εκτελείται διαφανώς. Λογοδοτήσει στο Ευρωκοινοβούλιο ήδη έχουν εκδοθεί πέντε εκθέσεις, τρεις ΕΣ και δύο για τέτοια και έχουν διατεθεί στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Να πω ότι τώρα που μιλάμε προχωρούν οι εργασίε. Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος για την εφαρμογή και των δύο συστημάτων. Και το σύστημα εισόδου-εξόδου αποτελείται από τέσσερα στοιχεία. Το σύστημα ΙΕΣ και ο οργανισμός ολοκληρώνει τις τεχνικές προδιαγραφές λεπτομερώς και η ανάπτυξη του συστήματος θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, το ίδιο ισχύει και για την εθνική ομοιόμορφη, ε, σημείο διαπαφής. Έχουμε το βιομετρικό σύστημα, ξεκίνησε, έχει προκυρηθεί ο διαγωνισμός και θα υπογραφούν οι συμβάσεις για την εφαρμογή του συστήματος το πρώτο τρίμηνο του 2020. Τρίτη συνιστόσα. Οι αλλαγές στο σύστημα πληροφοριών τη θεωρήσης που προέρχονται από το e από τον οργανισμό, έχει γίνει μελέτη αντικτύπου και ο οργανισμός ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις με τους συμβαλόμενους για το VIS για να ολοκληρωθούν οι διευθετήσεις και η υλοποίηση θα αρχίσει οι αρχές του 2020. Τέλος, εξής σημαντικό, η σημαντική συνιστόσα του ΙΕΣ e είναι το στο δίκτυο για τις πληροφορίες για τις θεωρήσεις. Προχωράει το έργο όπως είχε σχεδιαστεί και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Πέραν αυτού, οι διοικητικές δομές για το σύστημα ΙΕΣ, το σύστημα ε, διαχείρισης και διοίκησης και συμβουλευτική ομάδα που θα κατευθύνει επιχειρησιακά τις εργασίες και θα συντονίζει εργασίες μεταξύ κρατών μελών, οργανισμού και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύστημα εισόδου-εξόδου θα είναι θέσιμο για τα κράτη-μέλη να ξεκινήσει τη διαδικασία δοκιμών που είναι περίπλοκη διαδικασία το τέλος του 2020 και θα τεθεί σε ε, εφαρμογή το Φεβρουάριο του 2022. Αναμένεται ότι μετά σε θέση λειτουργία το σύστημα περίπου 400 εκατομμύρια συναλλαγές ε, το χρόνο θα εξετάζει εισόδου-εξόδου. σε περίπου 30.000 σημεία διέλευσης. Όσον αφορά το αιτίας, έχει σημειωθεί καλή πρόοδος. Ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία των αναγκαίων εφαρμοστικών πράξεων και κατεξοδότηση πράξεων. Προχωρά ε, το πρόγραμμα όσοι είχε σχεδιαστεί. Περιμένει ο οργανισμός όλες τις κατεξοδότηση πράξεις να είναι έτοιμες η εφαρμογή του συστήματος για να έχουμε το πρώτο τρίμηνο το κατάλληλο κείμενο και να προχωρήσουμε όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για το σύστημα. Παράλληλα, ο οργανισμός προοδεύει στον φάρο την προετοιμασία των διαγωνισμών. Εκεί θα συμπλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του κεντρικού συστήματος αιτία που πρέπει να αναπτυχθεί και, και, και διάφορες εφαρμογές, ε, ιστοσελίδα και τις γενικές υποδομές. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες και η ανάψη του, του συστήματος θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός προχωρά και με την πρόσληψη προσωπικού. Συγγνώμη, μας λένε ότι ίσως πρέπει να πάτε πιο σιγά για τους διερμηνείς. The same time, agency is progressing with recruitment of the... Προσλαμβάνουμε και άλλο προσωπικό, συμπληρωματικό προσωπικό, σύμφωνα με τον κανονισμό αιτίας. Για το αιτίας έχουμε και τις διάφορε διάφορες διοικητικές δομές, το Διοικητικό Συμβούλιο, Συμβουλευτική Ομάδα, για να συντονίζουν εργασίες μετά του οργανισμού κρατών μελών Frontex, Europol και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τετίας αναμένεται να λειτουργήσει τέλος του 2022, αλλά η εφαρμογή αιτίας και σύστημα εισόδου-εξόδου βλέπετε και από τη διαφάνεια ότι εντάσσεται σε ευρύτερη πρωτοβουλία για δηλετουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληροφορικής του συστήματος εσωτερικών και της αρχιτεκτονικής δομής του συστήματος πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαλειτουργικότητα έχουμε συνεργαστεί για το αιτίας σύστημα εισόδου εξόδου και είπα, εξετάζουμε διαλειτουργικότητα σύμφωνα με τον κανονισμό τον αρμόδιο. Η διαλειτουργικότητα μαζί με το αιτίας και το σύστημα εισόδου εξόδου θα εφαρμοστούν. Θα χρειαστούμε 9 με 12 μήνες για τη διαλειτουργικότητα. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το αίτιας και το σύστημα εισόδου-εξάδου είναι βασικά στοιχεία της διαλειτουργικότητας. Δεν έχουμε διαλειτουργικότητα αν δεν έχουμε τα άλλα δύο στοιχεία. Πιθανότατα, όπως βλέπετε από τη διαφάνεια, ότι η διαδικασία είναι περιπλοκότατη. Υπάρχουν εξαρτήσεις προβλήματα προς επίλυση. Ποια είναι τα πιο σημαντικά όσον αφορά τις εξαρτήσεις. Μεγάλη εξάρτηση από την έγκαιρη εφαρμογή του αίτιας και συστημάτων εσοδου εσόδου-εξόδου ε, εξαρτώνται από τις νομοθετικές διατάξεις. Κυρίως το Eurodac και ε, εφαρμοστικές διατάξεις. Άλλη εξάρτηση. το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε επαρκή χρήματα και επαρκές προσωπικό για να κάνουμε τη δουλειά μας. Την πρώτη διετία της νέας προγραμματικής περίοδου, τότε θα έχουμε τις σημαντικές εξελίξεις. Πρέπει να κάνουμε τι συμφωνίες, πρέπει να λειτουργήσουν τα συστήματα. Αυτό ήδη το θέσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Προεδρία. Για τα προβλήματα. Τρία είναι τα βασικά. Το πρώτο, συντονισμός, πολιτικός έλεγχος και προσανατολισμός για την εφαρμογή του συστήματος σε κεντρικό και εθνικό επίπεδο. Η εφαρμογή του αίτιας και του συστήματος εισόδου και εξόδου πρέπει να διευθετείται σε επίπεδο τεχνικό και λειτουργικό, επιχειρησιακό, αλλά σε πολιτικό. Το είπα στους Υπουργούς Εσωτερικών χτες στο Συμβούλιο, το αρμόδιο. Δεύτερο πρόβλημα πρέπει να δεχτούμε ότι η εφαρμογή των δύο συστημάτων εισόδου, εξόδου και δεν είναι τεχνικό πρόγραμμα. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στη δημιουργία δυνατοτήτων, στην κατάρτιση, διότι αν αυτόν δεν θα είναι αποτελεσματικά τα συστήματα. Το Ιουλίζα ήδη κατέβαλε μεγάλες σχετικές προσπάθειες μαζί με ΣΥΠΟΛ και Frontex και ετοιμάστηκαν προγράμματα κατάτησης για το EIS και για το ETIAS ε στα κράτη-μέλη και θα δώσουμε την κατάλληλη υποστήριξη αν χρειαστεί. Τρίτο πρόβλημα. Η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων. Η εφαρμογή επιτυχής των συστημάτων που συζητούμε εξαρτάται και από αεροδρόμια, ε, φορείς αεροδρομίων, ιδιωτικούς φορεί εν γέννη και πρέπει να το λάβουμε υπόψη στην εφαρμογή των συστημάτων που κουβεντιάζουμε. Και παρόμοιε πρωτοβουλίε έχουν εφαρμοστεί σε άλλε χώρε και τι παίρνουμε για προγράμματα. Το Ιλίζα εφαρμόζει, προχωράει για τη υλοποίηση των δύο προγραμμάτων. Έχουμε στενά χρονικά περιθώρια. Χρειάζεται συντονισμό σε κεντρικό και σε εθνικό επίπεδο. Το ΙΛΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για τα κεντρικά συστήματα να είναι έτοιμα εγκαίρω. Κοινή ευθύνη κρατών με, με τα κράτη-μέλη όμω ε, είναι η λύση για να πετύχουμε. Το ΙΛΙΖΑ συνεργάζεται στενά, επικοδομητικά με τα κράτη-μέλη, Frontex, Europol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουμε σωστά τα μέσα. Προσέχουμε ιδιαίτερα τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων. Θέλουμε τα νέα συστήματα να συμμορφώνονται απόλυτα. Τέλος, το Ελίζα θα παραμείνει σημαντικός εταίρος του Ευρωκοινοβουλίου για την υλοποίηση των συστημάτων. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να εξασφαλίσουμε έγκαιρη υλοποίηση σε κεντρικό επίπεδο και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κιόρκοφ για την πλήρη παρουσίασή σας, ειδικά για την Λίσσα. Ας ακούσουμε την έκθεση του κυρίου Ράμος, υποδιευθυντής των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Europol για την εφαρμογή του, υπεύθυνο κυρίως για την εφαρμογή του ETIAS. Ε Ποια είναι η κατάσταση Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. To appreciate very much this opportunity to, to debrief. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ενημερώσω ε, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αυτών των σημαντικών προγραμμάτων του συστήματος εισόδου-εξόδου και του ΕΤΙΑ στη Europol. Προχωράμε σε επόμενες διαφάνειες. Ποιος είναι ο ρόλος της Europol σε αυτά τα πολύ σημαντικά έργα. Όπως ξέρετε, ο καονισμός, ο σχετικός, προβλέπει ότι η Europol θα πρέπει να εφαρμόσει μία λύση, ούτω ώστε να προσφέρει πρόσβαση μέσω του, της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης Αναζήτησης ε, στην ενδιαφερόμενη κοινότητα. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίζουμε τον κίνδυνο από πρόσωπα που προέρχονται από το χώρο Σέγγεν. Η Europol επίσης θα υποφεληθεί από αυτά τα δύο σημαντικά έργα, δηλαδή οι εγκεκριμένοι αξιωματικοί της Europol θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων ε, στα πλαίσια αυτής της ε, πλατφόρμας διαλειτουργικότητας. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν οι διοκτικές αρχές να συνεργαστούν με τις αρχές προστασίας των συνόρων προς το συμφέρον των πολιτών για να διαχειριστούμε τα σύνορα και οι συνοριοφύλακες θα συνεργάζονται με τους αστυνομικούς ε, στα πλαίσια διαφόρων ερευνών ε, για προβλήματα που δημιουργούνται από τη μετανάστευση. Ε, η Europol έχει εξουσιοδότηση στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας, ούτως ώστε να βοηθήσει τους εγκεκριμένους αστυνομικούς για τον συνοριακό έλεγχο να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ε, βάσεις δεδομένων. Ε, γίνεται η αναζήτηση στα συστήματα της Europol. Εδώ βλέπετε την περιγραφή των συστημάτων, βλέπετε τη διεπαφή μέσω της διαπαφής θα υπάρχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων μας. Αυτό προβλέπεται να είναι έτοιμο το 2020. Παρ' όλα αυτά έχουμε ετοιμάσει ε, τη διαπαφή αυτή, ε, είναι έτοιμη και χαιρόμαστε που η προσπάθεια της Europol ε, για να υλοποιήσει την ατζέντα της διαλειτουργικότητας έδωσε αυτό το απτό αποτέλεσμα που είναι ακριβώς αυτή η διαπαφή η οποία θα μας εξασφαλίσει την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων μας. Είναι σαφές ότι όταν τελειώσουμε την, τις εφαρμοστικές πράξεις θα πρέπει να χτενίσουμε λιγάκι το εργαλείο αναζήτησης, αλλά αυτό δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο. Είναι έτοιμη η Europol για να αντιμετωπίσει και να υλοποιήσει αυτά τα σημαντικά προγράμματα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για την αρχιτεκτονική του συστήματος. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε αυτή την εικόνα. Θα ήθελα να σας πω όμως ποια είναι η συνεισφορά της Europol στην ατζέντα διαλειτουργικότητας. Με κόκκινο βλέπετε την διεπαφή αναζήτησης για τη Europol. Είναι το εργαλείο ούτω ώστε να υπάρξει η ολοκλήρωση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Αναζήτησης που είναι πάνω-πάνω και στα δεδομένα της Europol που είναι κάτω από την κόκκινη διαπαφή. Έτσι προβλέπουμε λοιπόν την ολοκλήρωση και ένταξη και αλληλεπίδραση όλων των συστημάτων. Οι εγκεκριμένοι αξιωματούχοι της Europol θα έχουν πρόσβαση μέσω της ε, δικτυακής πύλης αναζήτησης στα διάφορα συστήματα υπό το πλαίσιο της ατζέντα διαλειτουργικότητας. Σύστημα εισόδου-εξόδου, ΕΤΙΑΣ, ε, Γυροντάς, ΒΙΣ ε, και ΣΥΣΕΣ. Ε, σύστημα πληροφοριών Σέγγεν δηλαδή. Έχουμε ολοκληρώσει αυτό το τεχνικό εργαλείο, αλλά τώρα έχουμε άλλα στοιχεία τα οποία δουλεύουμε. Πέρυσι ο Διευθυντής εξασφάλισε τη σωστή διακυβέρνηση του συστήματος. Ο κ. Δεβόλφ αποφάσισε να ετοιμάσει ένα πρόγραμμα για τη διαλειτουργικότητα για να μετρήσουμε ε, στο, το κατά πόσο έχουμε όλους τους απαραίτητους πόρους για να τελεσφορήσει αυτό το σημαντικό project. Το Μάιο του 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Europol ενέκρινε το νοδικό χάρτη της Europol για την διαλειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά τι είναι αυτό. Ο Γενικός Οδικός Χάρτης Διαλειτουργικότητας που έχει διάφορες προθεσμίες και όπου εμπλέκεται και ο Ιγιου Λίσσα, αυτές, αυτά τα χρονοδιαγράμματα τα έχουμε ε, ενσωματώσει στη δική μας υπηρεσία, στο δικό μας οργανισμό, για να ε, είμαστε έτοιμοι στις διάφορες ε, προθεσμίες. Συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν στενά, με τη Frontex, με την Ίγιουλίσα ούτω ώστε αυτό το project διαλειτουργικότητας να είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς οι Κομισιόν και οι οργανισμοί, οι ενωσιακοί οργανισμοί συνεργάζονται για αυτά τα θέματα. Δίνουμε τεχνική βοήθεια ε, για τις διάφορες εφαρμοστικές και τεξουσιοδότηση πράξης που αφορούν το project αυτό. Επίσης προσπαθούμε να δώσουμε και τεχνικές λύσεις για να έχουμε τους απαραίτητους τεχνικούς πόρους και να μην υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ των τριών οργανισμών. Επίσης, για την επόμενη χρονιά ετοιμαζόμαστε ούτως ώστε όλη η υποδομή να είναι έτοιμη για να ε, μας επιτρέψει να διεκπεραιώνουμε όλες τις συναλλαγές που θα λάβουμε το 2020. Ποιες είναι οι προκλήσεις. Μας απασχολεί το θέμα της ε, τεχνικής υποδομής της ε, Europol. Χρειάστηκε να βαθμίσουμε την ε, υποδομή γιατί υπήρχαν δύο προβλήματα. Όλα τα συστήματα που αφορούν την ατζέντα της διαλειτουργικότητας είναι συστήματα που δουλεύουν πολύ εντατικά κάθε ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24 ώρο. Η Europol έχει καλά συστήματα για να δώσει πληροφορίες στα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ε, για να διατηρούμε επικυρωπημένα τα συστήματά μας. Δεύτερη πρόκληση. Τα συστήματά μας θα πρέπει να, να αναβαθμίζονται. Είναι θέμα κλίμακας. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ισχύ, ούτως ώστε όλα τα αιτήματα από τα άλλα συστήματα, ειδικά το, από το ΕΤΙΑΣ και το σύστημα εισόδου-εξόδου, να ε, τα διεκπεραιώνουμε εγκαίρως. Έπρεπε λοιπόν να αναβαθμίσουμε εντελώ την τρέχουσα υποδομή πληροφορικής. Σε ό,τι αφορά ε, το business process, ε, την επιχειρησιακή διαδικασία. Έπρεπε να ξαναδούμε πώς δουλεύει η Europol. Είναι θέμα του δουσού. Και επίσης είναι και θέμα συμμόρφωσης Εστιάζουμε κυρίως στο να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι, οι επιχειρησιακές διαδικασίες ε, σέβονται τον κανονισμό προστασίας δεδομένων και το νομικό πλαίσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και τέλος, είναι θέμα πόρων. Πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους πόρους, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε, ότι θα τελεσφορήσουν αυτά τα έργα. Εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας υποστηρίξει και πιστεύω ότι αν του χρόνου έχουμε τους απαραίτητους πόρους, ε, το 2020 δηλαδή, θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Θέλουμε και στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου να έχουμε τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Αυτά από πλευράς μου. Είμαι στη διάθεσή σας, εφόσον έχετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράμος. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τον τελευταίο προσκεκλημένο, πρωτού δώσουμε το λόγο στα μέλη, τα οποία μπορούν να σηκώσουν χέρια τις κάρτες τους ε, για να μπουν στο κατάλογο και να κάνουν ερωτήσει στους ομιλητές. Έχουμε λοιπόν ε, μαζί μας τον Φαμπρίς Λεζερή, εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, για να μας ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, καλημέρα σας. Όπως βλέπετε, είναι θέμα συνεργασίας της ομάδας. Έχουμε λοιπόν ε, την Delta ε, Home που παρουσιάζει για το γενικότερο πλαίσιο. Έχουμε την Ιουλίζα, την Ευρωπόλ και εμάς. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το σύστημα εισόδου-εξόδου. Είναι πραγματικά αποτελέσμα ομαδικής εργασίας και ε, η εμπειρία μας στην ε, Frontex ε, λέει ότι το μέλλον θα είναι στενά συνδεδεμένο με το σύστημα αυτό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι δραστηριότητε αυτές δεν έχουν να, κάνουμε με, να κάνουν με περιπτώσεις ε, κρίσεων, με παράτυπη μετανάστευση και με τα Είναι καθημερινές εργασίες μας. Στην Frontex, η, το στήσιμο όλο της κεντρικής ε, μονάδας του συστήματος ε, είναι δική μας λοιπόν αρμοδιότητα. Είναι ένα μέρος από ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από διάφορα συστατικά στοιχεία και εξού η διαλειτουργικότητα. Πρώτον, υπάρχει η κεντρική μονάδα του αίτιας που ε, πρέπει ακόμα να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί, αλλά έχουμε και ε, θέματα πρόσβασης στο SAS2 από την ακτοφυλακή και τη συνοριοφυλακή. Μετά, πρέπει να, να υλοποιήσουμε και ένα άλλο στοιχείο, το σύστημα δηλαδή υποβολής ε, εκθέσεων. Μετά έχουμε να κάνουμε με τη στήριξη των κρατών μελών ε, στην εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου. Εδώ θα επανέλθω. Δηλαδή το πώς εμείς ε, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για τους ελέγχους στα σύνορα και έπειτα είμαστε επιφορτισμένοι με, την, ε, με τον εντοπισμό ε, ατόμων που χρησιμοποιούν ε, πολλές ταυτότητες. Η κεντρική μονάδα λοιπόν είναι ένα σημαντικό στατικό στοιχείο, όμως δεν πρέπει να την εξετάζουμε μεμονωμένα, αλλά ως κομμάτι συνόλου. Το σύστημα αυτό το διαχειρίζεται ένα συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είμαι εγώ. Συνεδριάζουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και υποβάλλουμε εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ε, εφαρμογή τα στάδια του αίτιας. Και θα σας παρουσιάσω λοιπόν κάποιες από τις σημαντικότερες πτυχές ε, της ε, εφαρμογής. Πρώτον, η Frontex διοργανώνει σεμινάρια για τους εσωτερικούς συνεργάτες, για εμάς τους ίδιους δηλαδή, διότι η χρήση του συστήματος έχει άμεσες επιπτώσεις στη δουλειά μας. Και επίσης φροντίζουμε το σύστημα αυτό να είναι κατανοητό και ευρέως αντιληπτό, καθώς επίσης ε, και να γνωρίζουμε όλες τις επιτυχίε του σχετικού κανονισμού. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς είναι η ευθυγράμμιση των εργασιών με το σύστημα με την EU αλλά και με άλλους εταίρους. Επίσης, Προετοιμάζουμε το έδαφος για την πρόσληψη νέου προσωπικού που θα επανδρώσει την Task Force. Ξεκινήσαμε 1η Ιανουαρίου 2019. Και αυτή τη στιγμή καταρτίζουμε τον ορισμό και τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή την κεντρική μονάδα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εντοπίσουμε διάφορα σημεία γεωγραφικά στα οποία θα επεκταθούμε. Έχει να, πρώτον δηλαδή πρέπει να βρούμε την έδρα όπου θα ξεκινήσουν οι δοκιμές. Αυτό θα γίνει στη Βαρσοβία, δηλαδή στα κεντρικά του οργανισμού. Όμως, επειδή ο οργανισμός μας μεγαλώνει, θα πρέπει να αλλάξουμε έδρα και θα υπάρχει μία προσωρινή μονάδα όπου θα διχειρίζεται το αίτιας μέχρι να μετακομίσουμε στη, στα μόνιμα γραφεία μας. Έπειτα. Ασχολούμαστε και με θέματα σημαντικών υποδομών, με σχέδια έκτακτης ανάγκης. Εδώ συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Και επίσης ασχολούμαστε με τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Τώρα, για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει καταρχάς να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, έγκριση των ε, εκτελεστικών πράξεων και των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Στηρίζουμε την Λίζα με σημαντικές πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη. Από την πλευρά δηλαδή του χρήστη, εμείς συνεισφέρουμε και στην Ιουλίζα και στην Κομισιόν με τις γνώσεις μας. Στηρίζουμε όλο ένα και περισσότερο τα κράτη-μέλη με διάφορες ε, συναντήσεις έτσι ώστε να γνωριστούμε, έτσι ώστε να ενημερωθούμε. Συμμετέχει και η Ιουλίζα και η Ευρωπόλη σε αυτές τις συναντήσεις. Και αυτό γίνεται ακριβώς διότι το αίτια θα έχει άμεσες επιπτώσεις ε, στην καθημερινότητα των υπαλλήλων όλων αυτών των οργανισμών, αλλά και της συνοριοφυλακής. Έπειτα, συμμετέχουμε ενεργά στον ε, συντονισμό η Γιουλίζα, Ευρωπόλ και Frontex. Συνεδριάζουμε περίπου μια φορά το μήνα. Και Πρόσφατα εντοπίσαμε την ανάγκη να επεκταθούμε και στο σύστημα εισοδεξοδού και στο αίτιας και να ε, ξεκινήσουμε προκαταβολικά κάποιες ε, ενέργειες για τη σωστή χρήση τους. Πριν ξεκινήσει να λειτουργεί η κεντρική μονάδα του αίτιας. Φυσικά, όπως θα δείτε και στην έκθεσή μας, έχουμε εντοπίσει και κάποιους κινδύνους. Καταρχάς, με τα τεχνικά πρότυπα υπάρχουν κάποιοι νομικοί κίνδυνοι σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας. Επίσης, έχουμε διαπιστώσει θέματα πρόσληψης προσωπικού που θα στελεχώσει την κεντρική μονάδα. Εδώ υπάρχουν διάφορα λεπτά θέματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την έψο για τις προσλήψεις προσωπικού, διότι θα χρειαστεί να προσληφθούν περίπου 200 υπάλληλοι σε διάφορα στάδια. 250, με συγχωρείτε. Και θα χρειαστούμε λοιπόν τη στήριξη της ΕΠΣΟ για να το πράξουμε αυτό, έτσι ώστε να καταφέρουμε να το κάνουμε πρόθεσμα. Ε, πίτα. Πίτα, έχουμε εντοπίσει κινδύνους και με το Career Assistance Center. Θέλ, Έχουμε λοιπόν εντοπίσει διάφορα ζητήματα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας με τις αεροπορικές εταιρείε, με τους αερομεταφορείς. Γι' αυτό λοιπόν θα χρειαστεί να γίνουν και εκεί πολλά μέχρι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή έχουμε μία προσωρινή έδρα, θα ε, τη χρησιμοποιήσουμε μέχρι το Μάιο του 2021 Αναφέρομαι στην ε, προσωρινή έδρα την κεντρική μονάδα. Θα υπάρχουν δύο κύματα λειτουργίας, το πρώτο το 2021 και το δεύτερο το 2022. Αυτά ως προς τους ε, χειριστές υποθέσεων που θα δουλεύουν στο κέντρο αρρωγής για τις αεροπορικές εταιρείε. Αναμένεται να λειτουργήσουν όλες τι αρχές του 2022. Αυτά σε ό,τι αφορά την κεντρική μονάδα του αίτιας. Σας ε, μίλησα για το σύστημα εισόδου-εξόδου. Ο νομοθέτης όταν ενέκρινε τις σχετικές πράξεις δεν είχε υπόψη του τη Frontex το 2014 αυτό πολλά χρόνια πριν δηλαδή, αν συγκρίνουμε την νομοθεσία που είχαμε τότε με εκείνη που έχουμε τώρα. Μας προσκάλεσαν και άλλοι φορείς, η Γιουλίζα για παράδειγμα, να συμμετάσχουμε κι εμείς και δεχτήκαμε φυσικά. Παρέχουμε στήριξη στους συνοριοφύλακες από την ε, δική μας πλευρά και βλέπουμε ότι το σύστημα εισόδου-εξόδου και ύστερα το αίτιας ε, χαρακτηρίζονται από μεγάλη διασυνδεσιμότητα και θα αλλάξουν τον τρόπο που εργάζονται οι αρχές στα σύνορα. Θα χρειαστεί βέβαια εξυγχρονισμός, αλλά πρέπει να προετοιμάσουμε τη φυλακή για τις αλλαγές αυτές διότι το θέμα είναι να υπάρχει ένα σύγχρονο σύστημα σε λειτουργία. Αυτά σε ό,τι αφορά τις ε, νέες μας αρμοδιότητες, τη Frontex 2, το σύστημα που θα ξεκινήσει αύριο θα περιλαμβάνει πρόσθετες αρμοδιότητες και θα πρέπει μαζί με την ΣΥΠΟΛ και την Ιγιουλίζα να καταρτήσουμε το προσωπικό και φυσικά να τροποποιηθεί η εντολή μας ε, σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Επίσης έχουμε ξεκινήσει κάποια πιλωτικά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ή όπως και να έχει στην χρήση του συστήματος εισόδου-εξόδου από τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, θα πρέπει να το χρησιμοποιούν όλοι οι σταθμοί διέλευσης στα σύνορα. Και φυσικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε τη στήριξη που παρέχουμε σε περίπτωση που υπάρξουν δυσκολίες. Αν μπορούμε λοιπόν να στείλουμε κάποιο μόνιμο σώμα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Συμπερασματικά λοιπόν, έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Και όταν μιλάμε για την εντολή της Frontex, οι περισσότεροι ίσως θα έχουν κατά νου θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας. Όμως ε, θα ήθελα να πω ότι καλύπτουμε μεν θέματα παράτυπης μετανάστευσης και τους σχετικούς κινδύνους, καθώς και τους ε, κινδύνους που μπορούν να προκύψουν ε, σε θέματα ασφάλειας, για παράδειγμα από τους ξένους μαχητές. Όμως ε, το έργο μας αφορά και την ε, διευκόλυνση του ταξιδιού για τους καλόπιστους ταξιδιώτες. Κάθε χρόνο υπάρχουν πάνω από 600 εκατομμύρια νόμιμες διελεύσεις στα σύνορα. Οι περισσότερε από αυτέ γίνονται από πολίτε τη Ένωση. και αν συγκρίνουμε λοιπόν αυτά τα πάνω από 600 εκατομμύρια νόμιμες διελεύσεις με τις περίπου 150.000 παράνομες διελεύσεις, τότε θα δείτε ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε στη νόμιμη διέλευση, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους ε, πολίτες αλλά και να έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία, να είναι τα μεθορικά αυτά σημεία σε ετοιμότητα. Διότι μην ξεχνάμε ότι το ζητούμενο εδώ είναι η ομαλή διέλευση ανθρώπων και αγαθών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα τώρα. Ερωτήσεις. Τα μέλη να σηκώσουν το χέρι τους αν θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις, να σηκώσουν την κάρτα τους. Βλέπω το πρώτο χέρι να το σηκώνει κυρία Στίκ. Πρώτοι είσαστε εσεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους τέσσερις για αυτά που μας είπατε. Το όλο σύστημα συνεπάγεται και πολλές ανησυχίες δικές μας για τη θέματα ιδιωτικότητας, ορθότητα δεδομένων κλπ. Όταν κάτι πάει στραβά και τα συστήματα δεδομένων καμία στιγμή αποτυγχάνουν, υπάρχει και το θέμα των δικαιωμάτων των ιδιωτών. Η αρχή του περιορισμένου σκοπού δεν έχει αλλάξει. Πώς μπορεί να διαφυλαχθεί. Το όλο σύστημα συνεπάγεται περισσότερα δεδομένα για διαφορετικούς σκοπούς να είναι προσβάσιμα από διαφορετικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με διαφορετικά καθήκοντα. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η αρχή περιορισμένου σκοπού χρήσης των δεδομένων διαφυλάσσεται, τηρείται. Σχετικά με αυτό, έχουμε και τη ρήτρα περί μη διάκρισης και διατάξεις περί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το θέμα της διάκρισης. Φαντάζομαι ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι πληροφορίες περί αυτών είναι δυσανάλογα παρόντα στις βάσεις δεδομένων. Πώς να αποφύγουμε ότι έμεσα δεν θα υπάρχει διάκριση κατά αυτών των ανθρώπων. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναφερθεί σε αυτό. Πώς η διαδικασία υλοποίησεως εμπεριέχει μέτρα διαφύλαξης προς αποφυγή διάκρισης. η σημαντοδότηση, η ταυτοποίηση έχει δημιουργήσει ανησυχίες. Πώς είμαστε σίγουροι ότι κάποιοι που έχουν σημανθεί μπορούν να διαγράψουν τα στοιχεία τους, αν είναι λανθασμένα. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους όρους πρέπει να δώσει κατεξουσοδότηση πράξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αφαιθεί σε αυτό. Ποια κριτήρια θα είναι για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, Εποπτεία μετά και υλοποίηση. Εξαρτώμεθα σε μηχανισμούς εθνικούς εποπτείας και ξέρουμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί είναι περιορισμένοι. Και αυτά τα καθήκοντα που συζητούμε θα είναι πρόσθετα στα προβλεπόμενα τώρα. Άρα πώς θα μπορούν να εκτελούνται σωστά ε, αυτά τα καθήκοντα. Ευχαριστώ την ερώτησή σας. Η κυρία Κελέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Μας καθησυχάσατε. Συμπληρώσατε ένα στον άλλο με αυτά που μας είπατε. Ερωτήσεις τεχνικές και γενικές έχω. Κύριε Γκάρκοφ, ο πίνακάς σας ήταν άκρος ενδιαφέρον, αλλά δυσανάγνωστος. Οι πίνακές σας δυσανάγνωστοι. Το European Search Portal, αυτή η πύλη Αναζήτηση. Πώς λειτουργεί, τι είναι, περί τίνος πρόκειται. Οι εθνικές διοικησει θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή την πύλη για αναζήτηση. Και το Multiple Identity Detector, το σύστημα εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων, πώς λειτουργεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό από ό,τι κατάλαβα. Ο κύριος Σουλούν αναφέρθηκε 13 ε, κατεξοδότηση πράξεις, 16 εφαρμοστικές πράξεις, δεν έχουμε τίποτα να πούμε διότι είναι κατά εξουσιοδότηση. Κάποια στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε μια παρουσίαση περί προβλημάτων, περί προκλήσεων, περί δυσκολιών που χρήζουν προσοχής. Είπατε ότι στην κατεξουσιοδότηση προσέγγιση δεν ξέρετε αν θα είναι έτοιμα τα κάτι μέλη να εκτελέσουν μπορούμε να έχουμε κάποιες εξηγήσεις, να κατανοήσουμε την ολική. Κύριε Λεζερή, αναφερθήκατε στη συνεργασία με άλλες δομές που είναι παρούσες εδώ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάπως πώς αυτή η teamwork οργανώνεται, αυτή η μαδική εργασία, πώς οργανώνεται σε ευρωπαϊκή κλίμακα, αλλά και με τις διάφορες αρχές, τις εθνικές. Υπάρχει ε, διαχωρισμός, καθηκόντων, συντονισμός, πώς λειτουργεί. Άλλη ερώτηση. Αναφερθήκατε σε προβλήματα. Έχετε ένα σενάριο περί αντιμετωπίσεως κρίσεων. Είσαστε προετοιμασμένοι για μια κυβερνοεπίθεση Φερρυπίν. Κάποια συγκεκριμένη δυσκολία που θα καθιστούσε το σύστημά σας εύθραυστο. Ευχαριστώ. Κύριε Θοδωράτσι. ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω σαν τα βραβεία Όσκαρ, τα μέλη του πάνελ, που είναι όλα εδώ παρόντα. Είναι μια εικόνα διαλειτουργικότητας. Για πρώτη φορά βλέπω και τους τρεις φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ομιλούν αλληλοσυμπληρούμενοι περί των επιτευγμάτων. Είναι περίπλοκη η όλη διαδικασία. Σε ευχαριστώ που δίνεται μια εικόνα διαλειτουργικότητας. Τρει ερωτήσεις έχω. Πρώτη, ασφάλεια. Με τα συστήματα και πολλά σημεία πρόσβασης που δημιουργούνται. Θα έχουν πρόσβαση και συνοριοφύλακε σε κάποια συστήματα. Και μιλάμε και για δηλειτουργικότητα. Ανθρώπινο παράγων. Ο κίνδυνο από τον ανθρώπινο παράγοντα αυξάνεται όσον αφορά την ασφάλεια. Και εμεί που γνωρίζουμε κάπω πώ λειτουργούν τα συστήματα, ξέρουμε ότι ο ανθρώπινο παράγων καμιά φορά μπορεί να είναι πιο προβληματικό από τον τεχνολογικό παράγοντα όσον αφορά τους κινδύνους ασφαλείας. Πώς εξασφαλίζεται λοιπόν σωστό έλεγχο πρόσβασης και κωδικούς πρόσβασης για τους διάφορους αξιωματόχους των αρχών ε, των εθνικών, ε, συνοριοφυλάκων, αστυνομικών, ε, κοινοτικών φορέων κλπ. Και όσον αφορά την ασφάλεια. Συζητάμε τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Νέα στρατηγική που θα μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά διαχείριση δεδομένων. Τεχνολογία πέμπτη, πέμπτης γενιάς, 5G, δίκτυα ασφαλείας. Όλα είναι πολύ περίπλοκα όσον αφορά τα ψηφιακά και την ασφάλεια. Πώς θα εξασφαλίζετε ότι οι βασικές υποδομές και στοιχεία λογισμικού του συστήματος, για τον κύριο Γκάρκοφ είναι αυτό, στοιχεία λογισμικού λέγω, ελέγχονται και πιστοποιούνται σωστά όταν εισάγονται ως συνιστώσεις στο σύστημα. Είδα τις διαφάνειες που μας δείξατε και τα διαγράμματα. Είδα ότι είναι πολύ κομβική στιγμή για τους διαγωνισμούς για τα συστήματα τώρα. Άρα το θέμα της ασφαλείας των διαφόρων εξαρτημάτων και του εξοπλισμού είναι πρώτη στη μνά σα. Πώ εξασφαλείτε την ασφάλεια, μετά το χρονοδιάγραμμα. Βλέποντας τους πίνακές σας είδα ότι ήταν ε, περιπλοκότατο το εγχείρημα, με διάφορες συνιστώσεις διαλειτουργικότητας, παράλληλες εξελίξεις. Μέτρα ασφαλείας έχετε, ανάγκης στο σχεδιασμό. Πόσοι κίνδυνοι ελοχεύουν στο σχεδιασμό. Το ρωτάω αυτό, γιατί όπως ξέρετε συζητούμε και τα διάφορα στοιχεία που λείπουν από το νομοθετικό μείγμα, το VIS αίτιας, διαδοχικές τροποποίησεις. Εκεί το χρονοδιάγραμμα παίζει σημαντικό ρόλο. Για έκτακτες ανάγκες, τι μέτρα έχετε λάβει. Πόσο βασίζεστε στην ετοιμότητα των κρατών μελών να είναι έτοιμα όταν χρειάζεται και αν υπάρξει πρόβλημα πώς θα αντιμετωπιστεί όσον αφορά την ετοιμότητα. Μετά, κατάρτιση. Προετοιμασία όχι μόνο για του αξιωματούχου σα και ρωτάω και τον κύριο Λεζερή και την Europol αυτό, οι αξιωματούχοι των τριών υπηρεσιών που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα, πώ θα ετοιμαστούν, τι θα γίνει με την εκπαίδευση των αξιωματούχων των κρατών μελών που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Όταν κάνουμε διάφορες αποστολέ για το CIS και το VAIS και 10 χρόνια μετά την έναρξη των επιχειρήσεων υπάρχουν αρκετοί αξιωματούχοι των κρατών μελών που δεν γνωρίζουν πώ να χρησιμοποιούν σωστά τα υπάρχοντα συστήματα παρόλο που υπάρχουν για 10 χρόνια. Πώ θα προετοιμαστείτε για τη στιγμή που τα συστήματα αυτά που συζητούμε θα είναι έτοιμα, λειτουργικά, για να είμαστε σίγουροι ότι οι αξιωματούχοι των κρατών μελών θα είναι έτοιμοι να χρησιμοποιούν σωστά τα συστήματα. Ευχαριστώ. Κύριε Έρνστ, Ωραία, θα μιλήσω λοιπόν τη γλώσσα μου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη το ότι είμαστε 30 χρόνια μετά την πτώση του τείχου του Βερολίνου και γενικά όλων των ε, τυχών που χώριζαν Ανατολή ε, και Δύση και τώρα πάλι μιλάμε για δημιουργία άλλου τείχους ε, με, βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα κιόλα. Δεν το είχα, το φανταστώ εκείνη την εποχή. Και μου φαίνεται έτσι κάπως περίεργο όλο αυτό, σαν ένα δυσάρεστο ντεζαβού. Έχω μία δυσάρεστη παρατήρηση. Όπως γνωρίζετε, η δική μας ομάδα στηρίζει την διαλειτουργικότητα μεταξύ των αστυνομικών αρχών. Θεωρούμε πως είναι λογικό και πως πρέπει να ενισχυθεί για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Μην ξεχνάτε άλλωστε πως έχουμε ζήσει πολύ άσχημες στιγμές ε, τρομοκρατίας στην ε, Γερμανία. Όμως αυτή η σύνδεση που κάνετε της τρομοκρατίας με τη μετανάστευση είναι κάτι που μας βρίσκει ε, κάθετα αντίθετους και αρνούμαστε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια σύνδεσης αυτών των δύο. Μετά, Είπατε ότι η Κομισιόν, αν δεν κάνω λάθος, το είπε, ότι η συνοχή με τα άλλα συστήματα ε, έχει κάποιες εκκρεμότητες. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι εκκρεμότητες, τι παραμένει ανοιχτό, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των συστημάτων και τι πρέπει να γίνει ακόμα. Έπειτα, κάτι άλλο, ε, η κυρία Στρίκ το ανέφερε κιόλας, ε, σχετικά με την προστασία δεδομένων. Και έχω κι εγώ την ίδια ερώτηση. Θα ήθελα σας παρακαλώ λοιπόν να λάβατε θέση σχετικά με το πώς μπορεί να εγγυηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έπειτα, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά στάδια εφαρμογής, όπως ε, είπατε. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουν βελτιώσεις, όμως θα ήθελα να μας πείτε τι αναμένετε εσείς από τα κράτη-μέλη, τι εγγύσεις θέλετε να λάβετε, τι πρέπει να βελτιωθεί, ποια είναι τα αίτια των καθυστερήσεων και γιατί παρατηρούνται τόσο μεγάλες διαφορές ως προς ε, το στάδιο υλοποίησης. Και τέλος, για μένα πολύ σημαντικό, εσείς ε, θα ήθελα να μου πείτε το κόστος. Πόσο θα κοστίσει όλο αυτό το σύστημα από την αρχή μέχρι την εφαρμογή του. Πόσο θα κοστίσει η κατάρτιση προσωπικού, η πρόσληψη και τι κονδύλια διαθέτεται, τι δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι νομίζετε πως πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτά σε γενικές ε, γραμμές ε, και να πω ότι ε, έχω την εντύπωση πως τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να απομιστούν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μπράιν. Ευχαριστώ. Θέλω να τονίσω ότι είναι προβληματικές πολιτικές καταρχάς. Το σύστημα εισόδου-εξόδου συλλέγει αδιακρίτως στοιχεία από οποιονδήποτε ταξιδεύει. Ακόμα και μη υπόπτους. Δεν νομίζω ότι πληρούνται τα κριτήρια που έχει ε, θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη γνωμοδότηση για το PNR σε ό,τι αφορά το ETIAS. Ε ε, βάζουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιες πιθανότητες ε, με βάση α, ψευδείς αποκρίσεις, ε, false hits. Ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό, σωστές αυτές οι συνδέσεις. Σε ό,τι αφορά την έκθεση της Europol, α, που αναφέρει ένα-δύο ενδιαφέροντα σημεία. Καταρχάς λέτε ότι υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας για τις, σε σχέση με τις εθνικές βάσεις δεδομένων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιες είναι αυτές οι διαφορές και είπατε επίσης ότι η κρυπτογράφηση μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σίγουρο ότι αυτά τα δεδομένα θα κρυπτογραφηθούν. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι προφανές ότι θα πρέπει να κρυπτογραφηθούν. Τέλος, αναφέρατε το watch list, ε, το κατάλογο με πρόσωπα παρακολούθησης στα πλαίσια του ΕΤΙΑΣ. Ποιος θα μπει σε αυτό το κατάλογο, μια και τα κριτήρια είναι πολύ θολά, ασαφή για το ποιος θα μπορούσε στο μέλλον να διαπράξει ένα έγκλημα. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα στοιχεία για αυτό το πράγμα. Ο κύριος Λένερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχασα την αρχή της συζήτησης, λυπάμαι γι' αυτό. Δεν σκόπευα να πάρω το λόγο, αλλά μετά άκουσα ε, την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη αναζήτηση διάφορα πράγματα που με ενδιαφέρουν, εν πάση περιπτώσει, και τα έχουμε συζητήσει στο Κοινοβούλιο. Την πρώτη φορά που επισκέφθηκα επίσης το EU Λίσα, στο Στρασβούργο, ε, πήγα σε αυτό το υπόγειο, σε αυτή την, το μπούνκερ, ε, όπου είχαμε όλους αυτούς τους ε, σερβερ ε, που ήταν ο ένας εκατοστά από τον άλλον και όμως δεν επικοινωνούσαν γιατί είχαν διαφορετικούς πολιτικούς στόχους, ανήκαν σε διαφορετικές γενικές διευθύνσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και όταν τελειώσαμε ας πούμε τον γύρο αυτό και εξήγησα στο, στους ανθρώπους στο χωριό μου τι κάναμε, κανένα δεν μας είπε «Μπράβο σας», ε, αλλά μας είπαν, α, δεν φανταζόμουν ότι δεν τα είχατε ήδη στο παρελθόν ε, καταφέρει να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο και τώρα πάτε να το κάνετε. Ε, ο κόσμος πιστεύει ότι θα έπρεπε ήδη να είχαμε τη διαλειτουργικότητα ε, εξασφαλισμένη ανάμεσα σε αυτά τα συστήματα, ούτως ώστε να αυξήσουμε την ασφάλεια. Όταν μιλάτε για την ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ε, στη διαλειτουργικότητα ακριβώ ε, εξασφαλίζουμε αυτή την ισορροπία. Δεν αλλάζουμε τα δικαιώματα πρόσβαση, απλώ διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων και τα απαραίτητα τείχη. Και σε πολλού τομεί, χάρη στην ε, συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε βελτιώσει τι ασφαλιστικέ δικλείδε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων. Με μεγάλη χαρά άκουσα λοιπόν τα όσα είπαν διάφοροι και ο κύριο Τουντοράτσι και με χαρά βλέπω εδώ τους εκπροσώπους των διαφόρων οργανισμών εδώ μαζί είναι ένα σημαντικό μήνυμα ότι θα ξεφορτωθούμε αυτή την ε, προσέγγιση του κατακαιρματισμού σε ό,τι αφορά τις βάσεις δεδομένων. Και χαίρομαι που ακούω ότι η εφαρμογή προχωράει προς σωστή κατεύθυνση. Στο Κοινοβούλιο πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια και εμείς από πλευράς μας. Ορισμένοι ανέφεραν τις ε, τροποποίησεις που θα είναι η συνέπεια για το έτιάς. Ε την επόμενη Δευτέρα θα ακούσουμε την παρουσίαση στην, στην, εκπομπή... στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Αλλά δεν... και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους χρονικούς περιορισμούς. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας. Και μια τελική ερώτηση, ή μάλλον είναι η πρώτη ερώτηση, γιατί όλη την ώρα λέω παρατηρήσεις, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Πριν από καμιά δύο, εβδομάδε κάναμε συζητήσει για τα προβλήματα που είχαμε με τον προπολογισμό. Όχι το συνολικό ποσό, το συνολικό προπολογισμό, αλλά με τις προθεσμίες, ε, δηλαδή σε ποια φάση, σε ποια χρονική στιγμή εξασφαλίζουμε το τάδε επίπεδο ας και σε ποια χρονική στιγμή χρειάζεται μία υπηρεσία, ένας οργανισμός περισσότερα λεφτά από κάποιον άλλον. Κύριε Κέρκοφ. Αυτό εξακολουθεί να είναι πρόβλημα ή έχει επιληθεί στο μεταξύ. Αυτό ο συντονισμό, α πούμε, τη προθεσμία. Και για, στο μέλλον, για το προσωπικό. Ακούμε ότι είναι δύσκολο να έχουμε το κατάλληλο και επαρκέ προσωπικό. Όχι μόνο γιατί όταν αποφασίζουμε για το σύστημα εισόδου-εξόδου λέμε ότι αυτά τα άτομα ε, θα ασχολούνται με το σύστημα εισόδου-εξόδου και τα άλλα ε, άτομα θα ασχολούνται με το αιτιά, τα, τα, τα πούμε, άτομα θα ασχολούνται με τη λειτουργικότητα. Πόσο επηρεάζει αυτό τη λειτουργία των οργανισμών σας. Έχετε το επαρκές προσωπικό για να λειτουργήσουν οι οργανισμοί σας όπως πρέπει. Ευχαριστώ κύριε Λένες. Στάτλερ. Έχετε ερωτήσεις. Όχι, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, άρα παίρνουν το λόγο οι τέσσερις ομιλητές μας τρία λεφτά έκαστος, ούτω ώστε να μην καθυστερήσουμε και καθυστερήσει και το επόμενο σημείο. Ε, για το επόμενο σημείο, εξάλλου, βασικός ομιλητής είναι ο κύριος Λεζερή από τη Frontex. Ένας από τους τέσσερις πανελίστες μας εδώ. Επομένως, για να απαντήσουν οι ομιλητές με τη σειρά που μας έκαναν και τις αρχικές τους παρουσιάσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτές τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τρία λεπτά. Με δυσκολία, αλλά θα προσπαθήσω. Ε, δικαιώματα πρόσβασης, ε, περιορισμός, ποιος έχει πρόσβαση σε τι. Ε, για κάθε κανονισμό υπάρχει μια σαφής διάταξη που λέει για ποιο σκοπό η τάδε αρχή, ο τάδε φορέας έχει πρόσβαση στο σύστημα. Και το εφαρμόζουμε όλο αυτό με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να υπάρχει συνέπεια, κάθε τελικός χρήστη, κάθε φορέας να έχει πρόσβαση μόνο σε αυτό που του επιτρέπεται με βάση τον κανονισμό. Καθορίσουμε τα προφίλ των χρηστών που ισχύουν και για την διαλειτουργικότητα αλλά και για κάθε επιμέρου σύστημα και καθορίσουμε το προφίλ του χρήστη με βάση το περιεχόμενο του κανονισμού. Δεύτερον, ο τρόπος ε, πρόσβασης στο σύστημα καθορίζεται από την ανάγκη του να ξέρει. Ένα συνοριοφύλακα θα έχει πρόσβαση στο σύστημα με βάση το ταξιδιωτικό έγγραφο. Θα έχει το ταξιδιωτικό έγγραφο στα χέρια και μόνο με βάση αυτό το έγγραφο θα ρωτάει τα διάφορα συστήματα. Ενώ ένα άλλο χρήστη, α πούμε από τι διοκτικέ αρχέ, αστυνομικό κλπ, έχει άλλου τύπου πρόσβαση και έχει άλλε δυνατότητε να ψάξει ας πούμε, στο σύστημα και να αναζητήσει στοιχεία στο σύστημα. Επομένω, καθορίζεται και με ποιον τρόπο έχει πρόσβαση στο σύστημα ο κάθε χρήστη, ποιοι είναι οι περιορισμοί, τι δυνατότητε έχει να ρωτήσει και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες με βάση τη λειτουργία του κάθε φορέα, ας πούμε. Οι συνομοθέτες έχουν ε, συμπεριλάβει μια σειρά από διατάξεις και στο ε, και στο ΕΤΙΑΣ για να προστατεύσουν τα δεδομένα που υπάρχουν στο σύστημα και να δώσουν τη δυνατότητα στο φορέα να ζητήσει πρόσβαση για να ξέρει τι πληροφορίες έχει το σύστημα, να έχει το δικαίωμα αλλαγή, να, ε, να ρωτάει το σύστημα, δυνατότητα διαγραφής με βάση τις διατάξεις του κανονισμού, πάντα. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι τα συστήματα και τα βιοσυστήματα θα έχουν μια σειρά από εργαλεία τα οποία θα δοθούν στους ταξιδιώτες έτσι, στους επιβάτες, ούτως ώστε να γνωρίζουν την κατάσταση με βάση τα συστήματα, για να ξέρουν δηλαδή τι γίνεται ας πούμε με το σύστημα έγκρισης ε, του ΕΤΙΑΣ, να ξέρουν τον αριθμό ημερών που μπορούν να παραμείνουν στην επικράτειά μας, να ξέρουν πολύ καλά δηλαδή ποια είναι η κατάσταση και να γνωρίζουν πώς θα μπορούσαν να ταξιδέψουν ή να μην ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τους κανόνες για τη μέγιστη διάρκεια παραμονής. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τον ανθρώπινο παράγοντα που αναφέρθηκε από τον κύριο Τουντοράτσε, με το σύστημα εισόδου-εξόδου και το ΕΤΙΑΣ θα έχουμε μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της χρήσης από τον χρήστη. Αλληλεπιδρούμε με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή, ε, με τους χρήστες, το σύστημα με τους χρήστες, ειδικά με τους συνοριοφύλακες. Ε, η ανάγκη ε, ο συνοριοφύλακας επίσης να βάζει πληροφορίες καλύπτεται. Κάθε φορά που βάζει πληροφορίες, το σύστημα θα ρωτάει από το συνοριοφύλακα τι πρέπει να κάνει και θα τον καθοδηγεί για το πού θα βάζει τα στοιχεία. Ε, θα του λέει το άτομο αν μπορεί να μπει ή όχι. Και θα αφήσει βεβαίω την τελική απόφαση στον συνοριοφύλακα, αλλά θα του δώσει τι απαραίτητε πληροφορίε την κατάλληλη χρονική στιγμή. Θα τον βοηθήσει δηλαδή για να περιοριστεί και ο ανθρώπινος παράγοντας φάλματος. Ε, θα τον βοηθήσει το σύστημα το ίδιο δηλαδή. Για τον προϋπολογισμό. Απαραίτητο για τη λειτουργία των συστημάτων ή του συστήματος. Έχουμε μία νομική δημοσιονομική δήλωση που συνοδεύει τους δύο κανονισμούς και υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο ISF για να βελτιωθεί η κατάσταση στα χερσαία σύνορα και κυρίως στα σημεία διέλευση των χερσαίων σύνορων, ούτω ώστε να διευκολύνουμε αυτές τις χερσαίες ε, διελεύσεις. Έχουμε αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου στα σύνορα και χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατότητες μέσω των ε, τροπολογιών που έχουν υιοθετηθεί στον κώδικα συνόρων του Σέγγεν όταν ε, υιοθετήθηκε και το σύστημα εισόδου-εξόδου. Την ίδια χρονική στιγμή έγινε αυτή η αλλαγή δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα λέγω στον κύριο Γκάρκοφ για να αντιδράσει στα όσα ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω μέσα σε τρία λεπτά. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες στον κανονισμό οι οποίες εφαρμόζονται απόλυτα από τον οργανισμό μας στο πλαίσιο της χρήση του συστήματος εσόδου-εξόδου και ε, σε ό,τι αφορά το αίτια, επίσης υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης σε ισχύ. Τώρα, η κυρία Κέλλε ρώτησε για το ESP. Με λίγα λόγια, το σύστημα αυτό θα διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφορία. Θα κάνει δηλαδή όλα την αναζήτηση πιο αποτελεσματική, χωρίς να αποτελεί μια ανοιχτή πόρτα όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πάντες. Θα βοηθήσει τους ε, συνοριοφύλακες έτσι ώστε να έχουν γρηγορότερη, ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία. Επίσης, το, είναι ένα πάρα, το, ο εντοπισμό πολλαπλών ταυτοτήτων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι θα αποτρέψει αυτό το άτομο από το να χρησιμοποιεί διάφορες ταυτότητες για να εισέρχεται ε, σε έδαφο ένωσης, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν σε περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων. Επίσης, υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που χειρίζεται τα θέματα του συστήματος εισόδου-εξόδου και του αίτιας και εμείς έχουμε συντονιστικό ρόλο. Οι οργανισμοί Frontex και η Europol επίσης συμμετέχουν σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο και στις διαδικασίες ελέγχου. Τώρα, ε, φυσικά και παίρνουμε στα σοβαρά θέματα προετοιμασίας κυβέρνο ε, απειλής και τρομοκρατικού κυβερνοχτυπήματος. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τα κράτη-μέλη και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεκριμένες απαιτήσει και προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα κράτη-μέλη για τα τέτοια θέματα κυβερνοασφάλειας. Κύριε Τουντοράτσε, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, οι απαιτήσει ασφάλειας είναι ενσωματωμένες στις γενικότερες προδιαγραφές του συστήματος και επίσης ε, το ίδιο ισχύει για την πρόσβαση στην πληροφορία. Χρονοδιάγραμμα τώρα. Έχουμε αρκετά αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Ίσα ίσα μας παίρνει δηλαδή ο χρόνος μέχρι την θέση σε ισχύ και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τεχνικά ζητήματα αλλά και με πολιτικά. Ε, επίσης, Φυσικά και υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι στο θέμα της εφαρμογής, ιδιαίτερα από κάποια Όταν μάλιστα προσπαθεί σε κεντρικό επίπεδο να συντονίσει όλα αυτά, υπάρχουν δυσκολίε αν κάποιο κράτο μέλο δεν μπορεί να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα, γιατί πρέπει όλοι να περιμένουν μέχρι να είναι έτοιμο ο τελευταίο μαζί με την ΕΣΕΠΟΛ και την Frontex δηλαδή, συνεργαζόμαστε για να είναι όλα έτοιμα. Η πρώτη κατάρτιση θα γίνει το 2020 για να, για να καταρτιστούν οι χειριστές του συστήματος και μετά θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας δεδομένων, νομίζω πως ήδη ανέφερα ότι είναι ενσωματωμένα στον κανονισμό εφαρμογής εμείς έχουμε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προστασία δεδομένων. Οι βελτιώσεις που αναμένεται να κάνουν τα κράτη-μέλη έχει, να, έχει να κάνει με ε, όχι μόνο τεχνικά ζητήματα, αλλά με το πώς να ενσωματώσουν τις ε, νέες ικανότητες τις ήδη υπάρχουσες. Το σύστημα εισόδου-εξόδου και το σύστημα αίτιας λοιπόν θα προσθέσουν ικανότητες και πρέπει να ενσωματωθούν σωστά. Εμείς ε, φροντίζουμε να παρακολουθούμε αυτή τη σωστή ενσωμάτωση και των δύο συστημάτων και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και τον... για τον προπολογισμό. Όλα στηρίζονται στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Χρειάζεται προκαταβολή κάποιων κονδυλίων, front loading, αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν όλες, μέχρι να τελειοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες, ε, ακόμα βρισκόμαστε σε στάδιο διαπραγματεύσεων με τους συνομοθέτες. Έπειτα, ο οργανισμός μας ε, θα χρειαστεί κάποια επιπλέον ε, κονδύλια προς τη χρηματοδότηση από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για να μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του και για να εγγυηθεί τη διαλειτουργικότητα. Για παράδειγμα, το κόστος ε, της ε, σωστής λειτουργίας στο Στρασβούργο ανεβάζει τον προπολογισμό μας. Αυτά προς το παρόν από μένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάρκοφ. Κύριε Ράμος τώρα μπορείτε να συνοψίσετε ε, και εσείς σε λίγα λεπτά τις απαντήσεις ερωτήσεις των μελών. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω λοιπόν άμεσα σε ερωτήσεις σας σε ό,τι αφορά την διαπίστευση στην Ευρωπόλ. Εμείς αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε τρία διαφορετικά δίκτυα διαπίστευσης. Υπάρχει πρώτον η πρόσβαση στο σύστημά μας μέσω του επίπεδου βασικής προστασίας, όπως το ονομάζουμε, μέσω δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω των εμπιστευτικών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τρία επίπεδα διαπίστευσης δηλαδή. Ανάλογα με το είδος της πληροφορίας και το επίπεδο της ασφάλειας. Η πρόσβαση λοιπόν δίνεται στα κράτη-μέλη και σε τρίτους φορείς μέσω των τριών αυτών επιπέδων ε, διαπίστευσης. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα των ε, συστημάτων διαπίστευσης. Μπορώ να σας πω ότι αν για παράδειγμα ένα κράτος ε, μέλος έχει ένα βασικό επίπεδο προστασίας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να δίνει πρόσβαση σε αυτό το κράτος μέλος μόνο μέσω δικτύου VPN, VPL. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει αντιστοιχεία στα συστήματα που χρησιμοποιούνται και δεν θα πρέπει να δίνουμε πρόσβαση σε ένα κράτος μέλος αν για παράδειγμα υπάρχει ένα αίτημα από δίκτυο VPL για πληροφορία που κατατάσσεται σε εμπιστευτικό επίπεδο. Που χαρακτηρίζεται ως απόρριτη. Τώρα σε ό,τι αφορά αυτή τη watch Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή καταρτίζει τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Οπότε ίσως είναι πιο αρμόδια να απαντήσει αυτήν την ερώτηση, αλλά να σας πω ότι χρησιμοποιούμε συστήματα κρυπτογράφησης για τις απόρριτες πληροφορίες, ε, διπλής κρυπτογράφησης. Έτσι ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας για τις απόρριτες πληροφορίες. Όμως αυτά θα, περιλαμβάν, θα περιλαμβάνονται στις ε, εκτελεστικές και πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Και θα ακολουθήσουμε τις κατευθυντήσεις γραμμές που θα μας ε, δώσει η Κομισιόν. Τέλος, ε, το περιεχόμενο της πληροφορίας. Οι βάσεις δεδομένων θα πρέπει να περιέχουν το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο πληροφορίας. Θα πρέπει να είναι λοιπόν αποθηκευμένο ένα ελάχιστο επίπεδο στις βάσεις δεδομένων αλλά όχι στο watch Θα πρέπει να βοηθήσει δηλαδή τους συνοριοφύλακες και τις αστυνομικές αρχές ε, στις έρευνε τους. Αυτά λοιπόν πολύ σύντομα από μένα και ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λεζερή, η σειρά σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω γαλλιστή στην ερώτηση όσον αφορά το σχέδιο κρίσης όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Κάρκοφ. Προφανώς Υπάρχει ενίσχυση του συστήματος, των συστημάτων, έργο που γίνεται από την Ιγυλίζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν γέννη, εντός του οργανισμού μας ενισχύουμε το σύστημα πληροφοριών του Frontex και πέρα από το θέμα της κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με αυτά που θέλει ο νομοθέτης, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο για κρίσεις επεξεργαζόμεθα το θέμα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες υπηρεσίες το θέμα αυτό, το σχέδιο κρίσης, σχέδιο ανάγκης και είναι και θέμα φυσικής προστασίας των κτηρίων. Εξετάζουμε αν υπάρχει ανάγκη ή όχι να θεωρηθούν κρίσιμες υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή όσον αφορά το εθνικό επίπεδο όσον αφορά τη μονάδα αιτίας και τα σχετικά κτίρια πώς γίνεται η ομαδική δουλειά. Όχι μόνο συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών, αλλά μεταξύ κρατών μελών. Όπως καταλάβατε και όπως είπε και ο Κου, έχουμε ομάδες εργασίας τεχνικού επίπεδου, εκεί εκπροσωπείται τακτικά και η Frontex και άλλες υπηρεσίες, η Ιουλίζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συντονής Εργασίας και εκπροσωπείται τακτικά η Frontex Δημιουργήσαμε επίσης μία ομάδα υψηλού επίπεδου, ούτως ώστε να, να οι αρχές προστασίας των συνόρων συμπεριλαμβάνονται των κρατών μελών, που δεν έχουν αντιληφθεί ίσως τη σημασία του αιτίας και του συστήματος ε, entry-exit. Οπότε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η η Europol και τη Frontex τακτικά Δύο-τρεις φορές το χρόνο τα συναντόμαστε και εδώ και κάποιους μήνες άρχισα να δίνω ένα briefing στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ενημερώνω το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτά τα θέματα, ούτω ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να μπορεί να κατανοεί ακριβώ τι κάνουμε. Και αυτό είναι που επηρεάζει και τι εργασίε των εθνικών υπηρεσιών ελέγχου του ε, συνόλου. Και αυτό με φέρνει σε μία άλλη απάντηση. Δηλαδή, τι αναμένουμε εμείς από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, ε, υπάρχουν θέματα στα οποία ήταν ανεπαρκής η συμμετοχή της ε, συνοριοφυλακής ε, και των σχετικών αρχών. Θα πρέπει οι αρχές αυτές να είναι έτοιμες και καταρτισμένες ε, για την για τα νέα τους καθήκοντα, διότι τα συστήματα αυτά θα αλλάξουν τελείως τον ε, τρόπο λειτουργίας ε, του συστήματος, όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται κατάλληλη κατάρτιση. Και η τελική ερώτηση αφορούσε την κατάρτιση στα κράτη-μέλη. Βέβαιως θεωρούμε ότι είναι μια πρόκληση. Με το Ιουλίζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κατανοήσαμε για το σύστημα εισόδου-εξόδου. Θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή της υπηρεσίας όχι μόνο να εκπαιδεύσουμε τους δικούς μας συνοριοφύλακε, και εκεί θα έχουμε και άλλο πρόβλημα διότι θα έχουμε τα δικά μας μέλη του Ευρωπαϊκού Μονίμου Σώματος δεν μιλάμε μόνο για τα κράτη-μέλη και του αξιωματούχου των κρατών μελών και του συνοριοφύλακε των κρατών μελών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση ότι το προσωπικό κατηγορία 1 του μόνιμου Σώματος θα μπορεί να χρησιμοποιεί όλο τον εξοπλισμό τον τεχνολογικό Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους εθνικούς α, α, συναδέλφους μας στα σημεία ελέγχου των συνόρων, επιτόπου. Ευχαριστώ. Ξεπεράσαμε κατά πολύ το χρόνο στη διάθεσή μας, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Χαιρετίζουμε τα τρία μέλη του πάνελ, διότι έχουμε τον Φαμπρίς Λεζερή, που θα μιλήσει και στο επόμενο σημείο της ημίσης διάταξης, που θα αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή. Κάνα δύο λεπτά διάλειμμα να κάνουμε. Ένα λεπτό. <laughs> It'll be no time. Okay, now we go. Thank you, Monsieur Legeri, for your... Ο κ. Λεζερή, η μέρα σας είναι σήμερα. Παρακαλώ, αν παραμείνετε στην αίθουσα, να είστε ήσυχοι και αν αποχωρήσετε, να αποχωρήσετε ήσυχα, διότι έχουμε τη δουλειά μας, την ημερήσια διάταξη. Still a couple of time, a couple of points to go. A couple of points to go. Μένουν κανένα δύο σημεία. Για αυτό το σημείο είχαμε προβλέψει μία ώρα. Αλλά έχουμε μείνει πολύ πίσω. Ας συντομεύουμε λοιπόν αυτό το σημείο για να ακολουθήσουμε και με το άλλο. Αλλιώς θα έχουμε προβλήματα. This point concerns the implement... Εδώ μιλάμε για την εφαρμογή του θέματος των μέτρων για την Ευρωπαϊκή ε, Σύνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Ακόμα αποκαλείται Frontex. Άλλαξε όνομα όμως. Και στόχο. Και φύση. Και εμείς το κάναμε αυτό. Ανακατευθήκαμε, βάλαμε το χέρι μας σε αυτή την αλλαγή της Frontex που γίνεται η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Σημαντική νομοθεσία μας. Και γι' αυτό ευπρόσδεκτη ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με τον διευθυντή αυτού του γίγαντα, της γιγαντίας υπηρεσίας, του αστερισμού της ΛΥΜΠΕ. Νούμερο ένα, σε δυναμικότητα, προσωπικό, προϋπολογισμό και αυτό το πεδίο που καλύπτει μεταξύ όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την Επιτροπή μας. Ο Φαμπρίς Λεζερή θα παρουσιάσει εδώ τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το θέμα, με τον οργανισμό αυτό. Τον καλωσορίζουμε εκ νέου. Θα έχετε το λόγο. Τι σας προτείνω, σας προτείνω να προσπαθήσετε να μιλήσετε λιγότερο από ό,τι προβλεπόταν, για να έχουμε ακόμα περιθώριο ερωταπαντήσεων και να έχουμε και κάποιο χρόνο ή δυνατόν ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μερίσια διάταξη για σήμερα, που ακόμα έχει άλλο ένα σημείο. Έχετε το λόγο, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Όπω γνωρίζετε, η νέα εντολή, ο νέος κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα τεθεί σε ισχύ αύριο. όπω ξέρετε, ήδη ξεκινήσαμε την προετοιμασία κυρίως την ανάπτυξη του βασικού ευρωπαϊκού σώματος από 1η Πρώτου 2021. Θα θυμόσαστε ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνήσαμε επί οδικού χάρτη κοινού. Περιγράφονται τα καθήκοντα εκεί, το τι πρέπει να γίνει, πότε και ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Υπάρχουν και κάποιες επιτροπές βέβαια υπό την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για εφαρμοστικά μέτρα που πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντού. Να πω ότι πρέπει να εστιαστώ επί των σημαντικότερων δράσεων που ολοκληρώθηκαν. Πρώτα απ' όλα, από φέτος το καλοκαίρι κουβεντιάσαμε τις εθνικές υπηρεσίες, κυρίως με τους διοικητές των σύνοριοφυλάκων και των διαφόρων αρμοδίων αρχών που ασχολούνται με τη διαχείριση των σύνορων χερσαίων, θαλασσίων, εναερίων. Είναι κρίσιμο από κοινού να πετύχουμε το στόχο, όχι μόνο σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και με τα κράτη-μέλη. Μιλάμε για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και α, ακτοφυλακή που αποτελείται από τις εθνικές υπηρεσίες της αρμόδιες και τη δική μας υπηρεσία. Είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Είναι κάτι παραπάνω από μία έννοια. Είναι μία πραγματικότητα. Επεξεργαστήκαμε και νέα επιχειρησιακή έννοια Δηλαδή, πώς θα χρησιμοποιούμε το μόνιμο σώμα. Επεξεργαζόμαστε έναν κατάλογο υπηρεσιών που θα μπορεί να παραδίδει υπηρεσία στα κράτη-μέλη. Υπηρεσίες ποικίλουν. Από υποστήριξη στα σημεία διέλευσης, στα σύνορα, υποστήριξη για υποπτήρια των σύνορων, στήριξη για δραστηριότητες επιστροφής με δυνατότητες που θα αυξηθούν όσον αφορά την επιστροφή και εκούσια επιστροφή και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, μεγαλύτερη ανάπτυξη προσωπικού και δυνατότητες ανάπτυξης προσωπικού και δυνάμεων σε τρίτες χώρες. Αυτό που είναι σημαντικό βραχυπρόθεσμα είναι να ολοκληρωθεί η εκστρατεία προσλήψεων επιτυχώς. Η πρώτη φάση προσλήψεων ξεκίνησε τον Οκτώβριο. 23 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε, δημοσιεύθηκαν οι κενές θέσεις για το πρώτο κύμα προσλήψεων. 700 με 800 συνοριοφύλακες αναμένεται να προσληφθούν μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Προθεσμία για τις αιτήσει είναι 16 Δεκεμβρίου. Οπότε εργαζόμαστε σκληρά για να συνεργαστούμε με επαγγελματική εταιρεία για αυτά τα θέματα, για να κοινοποιηθούν σωστά οι πληροφορίες. Επιμένουμε στο ποιοτικό στοιχείο. Αυτό είναι απαραίτητο για εμπιστοσύνη η ποιότητα. Διότι τα κράτη-μέλη πρέπει να μας εμπιστευτούν, να γνωρίζουν ότι προσλαμβάνουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στο μόνιμο σώμα. Οι πολίτες πρέπει να μας εμπιστευτούν ότι έχουμε την κατάλληλη στελέχωση σωστοί άνθρωποι με την κατάλληλη εκπαίδευση που θα δίνουν αποτελέσματα. Η κατάρτιση θα διαρκέσει ένα εξάμεινο. Θα ξεκινήσει 1η Μαΐου του χρόνου η κατάρτιση μέχρι τέλος του έτους και σταδιακά θα αρχίσει η ανάπτυξη του σώματος από 1η Πρώτου 2021. Να πω επίσης ότι πλησιάζει η έγκριση των επαγγελματικών προδιαγραφών για τις θέσεις για τους συνοριοφύλακες που θα προσληφθούν τι καθήκοντα θα εκτελούν. συνοριακό έγκλημα, παραδείγματο χάρη, ακτοφυλακή, υπεύθυνο για επιστροφή, για έλεγχο των συνόρων, ειδικό για ανάλυση κινδύνου, Φερρυπίν. Διάφορε ειδικότητε, διότι όταν λέμε συνοριοφύλακα, αυτό δεν είναι αρκετά συγκεκριμένο όρο, γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτέ τι ειδικότητε. Σε κάθε δουλειά χρειάζονται ειδικέ ικανότητε και γνώσεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συμφωνήσουμε τα κράτη-μέλη στο επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης έχουμε προετοιμάσει τη νέα μεθοδολογία αξιολόγησης που θα είναι έτοιμη από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός για να ξέρουμε και ποιοι θα είναι οι διαθέσιμοι άνθρωποι. Έτσι θα ενισχύσουμε περαιτέρω το συσχετισμό με το σύστημα αξιολόγησης Σέγγεν και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάναμε πρώτες προετοιμασίες για το μοντέλο ανάπτυξης των αξιωματούχων αυτών και λεπτομέρειες πώς θα τοποθετηθούν. Πρέπει να σκεφτούμε ότι θα έχουμε ένα μόνιμο ευρωπαϊκό τέτοιο σώμα, δηλαδή μετακινούμεθα από το προηγούμενο σύστημα τοποθέτησης που ήταν τοποθέτηση ατόμων που διέθεταν τα κράτη-μέλη, τώρα θα έχουμε μεγάλες ομάδες ατόμων που βεβαίως θα συνεπάγεται και κάποια επιμελητία από τον οργανισμό. Αν τοποθετούμε χιλιάδες συνοριοφύλακες ή μέλη της ακτοφυλακής, δεν μιλάμε πλέον για άτομα που ψάχνουν να βρουν ξενοδοχείο κάπου για να στεγαστούν και μόνο πρέπει να προβλεφθεί η οργάνωση. Αυτό είναι το επιχειρησιακό μοντέλο και οι λεπτομέρειες ανάπτυξης αυτών των δυνάμεων και θα σωστή προσέγγιση θα επιτρέψει και οικονομίες. Αυτό είναι σημαντικό πλευράς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω επίσης ότι επεξεργαζόμαστε και τη μελλοντική στολή. Θα θυμόσαστε ότι το προσωπικό κατηγορίας 1 οι αξιωματούχοι τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για πρώτη φορά στην ιστορία θα φοράνε ευρωπαϊκή στολή. Έχουμε τα πρώτα σκίτσα για τη στολή. Πρέπει να κάνουμε πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής πριν υποβάλουμε τη στολή στο Διοικητικό Συμβούλιο μας. Συλλέγουμε λοιπόν εμπειρογνώμονες για όπλα, για εξοπλισμό, Ξέρουμε ότι η χρήση όπλων είναι κάτι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Ευαίσθητο καταρχάς για λόγους νομικούς, όπως καταλαβαίνετε το νομικό καθεστώς είναι περίπλοκο, διαφέρει σε κάθε χώρα που θα πηγαίνουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει σωστή συνεννόηση από αυτού. Πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Την κινητικότητα, των μέλων την κινητικότητα των μελών του μονίμου σώματος και πώς θα μεταφέρονται και τα όπλα του μονίμου σώματος. Συλλέγουμε εμπειρογνώμονες για αυτό το σκοπό και θέλουμε να έχουμε τις βέλτιστες προδιαγραφές και, τα... και τις βέλτιστες πρακτικές. Ο κανονισμός στελέχος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπει πρότυπα γι' αυτό. Δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για την ώρα εξοπλισμένοι που πλοφορούν. Είμαστε με την DH ε, ανθρωπίνων πόρων, HR, σε επαφή για να εντοπίσουμε τις λύσεις, να καθορίσουμε πρότυπα και προδιαγραφές όπου χρειάζονται εφαρμοστικά μέτρα, παραδείγματο χάρη. Ψυχολογικές δοκιμές, τεστ απαιτούνται και το προβλέψαμε αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε αξιωματούχους επιβολής του νόμου που δεν περνάνε από συνηθισμένες ψυχολογικές δοκιμασίες που είναι πολύ κοινέ στα κράτη-μέλη. Πρέπει να προσαρμοστούμε δεόντως ούτως ώστε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο είναι ιστορικής αξίας. Και η απόφαση του Ευρωπαίου νομοθέτη ήταν επίσης ιστορική. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν. Εδώ είμαστε. Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Ίσως ήταν καλύτερα να ολοκληρώσω εδώ, λέγοντας ότι είμαστε εντός των προθεσμιών, είναι στενές οι χρονικές προθεσμίες αλλά δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε όσον αφορά την υλοποίηση των σχεδίων. Ευχαριστώ τον Διευθυντή, τον κύριο Λεζερή, για την παρουσίαση. Point and Ο οποίο ήταν πολύ λακωνικός, άρα μας δίνει χρόνο για ερωτήσεις. Η κυρία Στάτλερ έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Μία λειτουργική ακτοφυλακή και ιστοριακή είναι προπόθεση για να λειτουργεί σωστά το Σέγγεν. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να μιλάμε για το θέμα αυτό και να τονίζουμε τη σημασία του. Δύο θέματα είναι σημαντικά και πρέπει να έχει την απαραίτητη εντολή η Frontex. Πρέπει να έχει τα απαραίτητα νούμερα και την κατάλληλη ποιότητα. Είπατε ότι τα άτομα αυτά χρειάζονται έξι μήνες κατάρτιση. Γίνεται και η πρώτη εκστρατεία ε, προσλήψεων μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου τρέχει η προθεσμία. Η Ursula von der Leyen ε, ζήτησε, έχει θέσει ως στόχο 10.000 άτομα στη Frontex ε, μέχρι το 2024. Ε, προηγουμένως η ημερομηνία ήταν 2027. Κάπως καλύτερα είναι, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ μακριά η προθεσμία δεδομένων των αναγκών που πρέπει να καλύψει η Frontex. Ε, σε αυτή την πρώτη εκστρατεία προσλήψεων μέχρι το Δεκέμβριο, πόσους θα προσλάβετε, ούτω ώστε να ξέρουμε πώ θα είναι έτοιμοι το επόμενο εξάμεινο. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, έχετε ένα σαφέ σχέδιο για αυτά τα 10.000 άτομα. Πόσα από αυτά θα σταλούν στα κράτη-μέλη και πόσα πόσα θα προσλάβουν μάλλον τα κράτη-μέλη και πόσα θα προσλάβει η Frontex. Είναι σημαντικό να το ξέρουν τα κράτη-μέλη. Επιπλέον το σώμα αυτό θα διαιρεθεί μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, έτσι δεν θα πάνε όλοι σε ένα κράτος μέλος. Κυρία Κέλλερ, μετά από τις προηγούμενες ερωτήσεις που ακούσαμε, συνεχίζω και εγώ με τις εξή. Για την πρόσληψη των ακτοφυλάκων και των σύνοριοφυλάκων, ε, πού θα ασκούν τα καθήκοντά τους πρώτον. οι οργανισμοί θα είναι τακτικά σε ορισμένου τόπους, σε ορισμένες περιοχές, ε, πόσοι θα είναι και πόσοι θα αποσπώνται, θα πηγαίνουν σε περίπτωση κρίσης. Ε, υπάρχει και η ποσόστοση των 10.000 ακτοφυλάκων ε, συνοριοφυλάκων, αλλά με ποιο ρυθμό θα προσληφθούν. Με τι συχνότητα θα προσλαμβάνετε άτομα. Με κυρία Βόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση και για τη δουλειά που έχετε κάνει. Θα μπω κατευθείαν στο ζητούμενο. Η Frontex λοιπόν έχει, μία, έχει ξεκάθαρες αρμοδιότητες με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει λοιπόν από τη μία αρμοδιότητα προστασία των συνόρων. Από την άλλη όμως οφείλεται να σέβεστε και τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την διαφύλαξη αυτή των συνόρων. Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του προσωπικού, σε ποιο σημείο βρίσκεστε και ποιε είναι οι ικανότητες που χρειάζονται έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να τηρήσει και τα δύο, διότι υπάρχουν διάφορα ε, προβλήματα και σε περίπτωση που συνεχιστεί προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι υπεύθυνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Στρίκ. Ευχαριστώ τον κύριο Λεζερή. Η ερώτησή μου ε, είναι η συνέχεια της ερώτησης των σοσιαλιστών σχετικά με την θέση του αξιωματούχου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, είναι ένα τομέα πολιτικής λίγο αβέβαιος. Υπάρχουν ε, έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι υπάρχουν παρατυπίες στα εξωτερικά σύνορα. Υπάρχει ανεξάρτητη παρακολούθηση από άτομα τα οποία έχουν πραγματογνωμοσύνη για το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο, μια και είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς πρόσβαση στο σωστό σημείο, ας πούμε, και να είναι υπάρχει διαφάνεια για το τι συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, στα διάφορα σημεία των σύνορων. Μια άλλη ερώτηση υπάρχει μια θέση που χειρεύει στην Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, και αυτό μας εντυπωσιάζει, γιατί ε, κανονικά υπάρχει πραγματογνωμοσύνη ε, από αυτή την, αυτό το άτομο που τώρα κατέχει αυτή τη θέση στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ξέρει πολλά πράγματα, υπάρχει, είμαστε σίγουροι για την εξαρτησία της κτλ. Τα έχει τονίσει αυτά το Κοινοβούλιο και το παλιό και το καινούριο και τώρα σε μια χρονική στιγμή που α, μεγαλώνει η Frontex, και υπάρχουν εκεί οι παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία που έχει ήδη ο αξιωματικός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί τώρα, αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η Frontex αποφασίσει να διώξει την, το άτομο αυτό και να προσλάβει ένα καινούριο. Γιατί χειρεύει αυτή, γιατί υπάρχει αυτό το κενό. Επίσης, τι σημασία δίνεται σε αυτό που εμείς τονίσαμε ως σημαντικό για την ανεξαρτησία και την πραγματογνωμοσύνη και για τη διαδικασία. Ο διευθυντής της Frontex παίζει μεγάλο ρόλο στην διαδικασία πρόσληψης ε, αυτού του αξιωματούχου της ε, Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω του πόσο σημασία δίνουμε στην ανεξαρτησία. Η Frontex ετοιμάζει ένα shortlist. shortlist Επίσης, το συμβουλευτικό φόρουμ, τι, σημαντικό, ε, τι ρόλο παίζει, ο κανονισμός προβλέπει σημαντικό ρόλο γι' αυτό, αλλά πώς τον παίζει αυτό το ρόλο. Επίσης, η πρόσληψη των παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό. Πρέπει να παρακολουθήσουμε πολλά πράγματα σε πολλά μέτωπα. Ε, στον δικό χάρτη της Frontex βλέπουμε ότι προβλέπεται να γίνει στα τέλη του επόμενου έτους. Γιατί να μην ξεκινήσει τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή. Ευχαριστώ που θέτετε αυτό το θέμα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τον αξιωματούχο και παρατηρητή θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εγώ θα το έθετα αυτό σε ερώτημα. Να προσθέσω και κάτι άλλο, μια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν εκπροσωπείται στην αίθουσα. Θα ήθελα να ακούσω όμως την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη τρέχουσα διαδικασία ε, και το κενό που υπάρχει στη θέση. Συνήθως είναι στην αίθουσα η Κομισιόν. Δεν είναι, δεν, δεν εκπροσωπείται. Αν δεν εκπροσωπείται, λυπάμαι. Βλέπω τα έδρανα της Κομισιόν. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να μιλήσει. Αν δεν είσαστε, να εκπροσωπήσετε πλήρω όπω πρέπει για να απαντήσετε τώρα, κρατήστε σημειώσει για να μα απαντήσετε. Γιατί το θέμα είναι σημαντικό. Θα το έθετα κι εγώ. Mr. your floor. Ο κύριο Τουντοράτσι, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ. Κύριε Λιζερή, καταρχάς σας ευχαριστώ για τον ε, οδικό χάρτη. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικός, πολύτιμος θα έλεγα, όχι μόνο από επιχειρησιακής πλευράς αλλά και για την εξέλιξη της Frontex, το, κάτι το οποίο είναι και ένα πολιτικό μήνυμα. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω να έρχεστε τακτικά και να μας ενημερώνετε καθώς ε, και για τις εξελίξεις της ε, ομάδας για το Σέγγεν. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε και εμείς ενημερωμένοι για την πρόοδο του οδικού χάρτη. Τώρα μας μιλήσατε για προσωπικό, για νέες προσλήψεις ε, και ε, νομίζω πως είναι πολύ καλό ότι καταφέρατε να πείσατε την ΕΠΣΟ να συμμετάσχει στην πρόσληψη νέου προσωπικού. Γιατί όντως θα χρειαστείτε αρκετούς. Έχω όμως μία ερώτηση σχετικά με ε, τους ε, Τι γίνεται με τον προϋπολογισμό σας, διότι καθώς βρισκόμαστε σε μία νέα περίοδο είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται στα οικονομικά. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα επιχειρησιακά κέντρα, είναι αυτό κάτι το οποίο εξετάζεται ως κομμάτι του οδικού χάρτη. Υπάρχουν συγκεκριμένες τοποθεσίες που προβλέπονται ε, να λειτουργήσουν αυτά τα κέντρα. Και επίσης τα περιουσιακά σας ε, στοιχεία. Από τη στιγμή που ξεκινάτε να αγοράζετε διάφορα σκάφη, που πούμε, ελικόπτερα, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα διαχείρισής τους. Ευχαριστώ πολύ. Αν κατάλαβα καλά, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Επομένως, κύριε Λεζερή, μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. It's uh, related questions. First of... Θα ξεκινήσω πρώτα με τις ερωτήσεις που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, το μόνιμο προσωπικό φυσικά και θα είναι παρκώς καταρακτισμένο, έτσι ώστε να έχει επίγνωση και να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την προκήρυξη για την ε, πλήρωση της θέσης ε, του υπεύθυνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτή τη στιγμή υπάρχει αναπληρωτής Και όπως είπατε και εσείς πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειες έτσι ώστε να προσληφθούν 40 τέτοιοι επόπτες θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έτσι ώστε να βρίσκονται στο πεδίο και να παρακολουθούν τη δράση μας. Νομίζω ότι αυτό συζητήθηκε στην Επιτροπή σας πριν τις ε, εκλογές. Και τώρα, έχουν συζητηθεί και τα θέματα ανάγκης αναβάθμισης, ε, πως ε, χρειαζόμαστε νέο προσωπικό, χρειαζόμαστε από το 2015 ε, τόσο προσωπικό όσο και περισσότερη χρηματοδότηση και βλέπουμε ότι τώρα ξεκινάμε μία άλλη φάση της λειτουργίας μας. Θα έχουμε πάνω από 10.000 μόνιμο προσωπικό. Αποφάσισε λοιπόν ο νομοθέτης ότι οι 40 επόπτες θα δίνουν αφορά μόνο στον ε, υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όμως, για να λειτουργήσει σωστά η ιδιότητα του υπεύθυνου θεμελιωδών δικαιωμάτων θα χρειαστεί και ένας ε, υπάλληλο με διευθυντικέ ικανότητες, κάτι το οποίο δεν έχουμε προς το παρόν. Γι' αυτό και έχουμε συστήσει να αναβαθμιστεί ο ρόλος αυτός, έτσι ώστε αυτή η θέση να ανήκει σε ανώτερη βαθμίδα, σε διευθυντική βαθμίδα και σύμφωνα με τον οδικό χάρτη θα πρέπει να υποβάλουμε μία πρόταση για τον αναπληρωτή υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα πρέπει δηλαδή να επιταχύνουμε εδώ και φυσικά να ξεκινήσουμε τη διαδικασία πρόσληψης των 40 υπαλλήλων που θα έχουν το ρόλο του επόπτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να υπάρχει ένας υπάλληλο που να έχει την κατάλληλη βαθμίδα, να ε, είναι σε αυτή την διευθυντική θέση που όπως γνωρίζετε δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, διότι οι θέσεις μας ε, δεν είναι τέτοιας βαθμίδας. Και ο λόγος που χρειάζεται να αναβαθμιστούμε είναι επειδή πρέπει να αναβαθμιστούν και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε. Και οι νέες ε, υπηρεσίες ε, που θα έχουμε στο μέλλον μέσω του, των αποπτών και του υπεύθυνου θεμελιδών δικαιωμάτων. Συν άλλοι 10 υπάλληλοι που έχουμε προς το παρόν που εργάζονται στο Γραφείο Θεμελιδών ε, Δικαιωμάτων, δηλαδή σύνολο 50 και δεδομένου του μεγέθους των μονάδων, αυτή η θέση σίγουρα θα πρέπει να είναι διευθυντική. Έχουν περάσει εποχές όπου ο υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων είχε έναν βοηθό και έναν ασκούμενο. Τώρα έχουν αλλάξει και οι τάξη, και μεγέθους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης των 40 εποπτών και να πω ότι επιπλέον έχω ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα με την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Όπως είδατε και από την παρουσίαση για το ΕΤΙΑΣ, για την Ευρωπόλη, συνεργαζόμαστε στενά με αυτούς τους ε, οργανισμούς και το ίδιο συμβαίνει και με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο τελεστικός διευθυντής της ΕΦΡΑ έχει υπογράψει μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών μας και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε συνεργασία μαζί μας έχει ξεκινήσει λοιπόν την εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος το οποίο αφορά έρευνα και επισκέψεις επιτόπου σε ορισμένα κράτη-μέλη που έχουμε προτείνει αμφότεροι για να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα, ένα πλαίσιο για τους 40 ε, αυτούς επόπτες. με το σκεπτικό να δημιουργηθούν κάποιες ε, κατευθυντήριε γραμμέ για αυτού τους επόπτες. Αυτή είναι η δική μου δουλειά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ Frontex και FRA σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το Μάρτιο, που ελπίζω να έχουμε και τις ε, πρώτες συστάσεις. Το Μάρτιο του 2020. και τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής θα τα χρησιμοποιήσουμε για την πρόσληψη του νέου προσωπικού ε, και των εποπτών και του μόνιμου σώματος. Δηλαδή θα τρέχουν παράλληλα και η πρόσληψη κατάρτιση προσωπικού και η κατάρτιση μέσω του πιλωτικού προγράμματος, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στο χρονοδιάγραμμα. 1η δηλαδή Ιανουαρίου 2021. που τότε αναμένεται να έχουμε ήδη στείλει τους πρώτους επόπτες στο πεδίο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, αν δεν κάνω λάθος με ρωτήσατε για την ε, αναλογία προσωπικού κατηγορίας 1 των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή και του ε, προσωπικού από τα κράτη-μέλη. Το 70% λοιπόν του προσωπικού θα προέρχεται από τα κράτη-μέλη και το 30% από τον ε, οργανισμό μας, από την κατηγορία 1. Αυτό σημαίνει ότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα υπάρχουν περίπου 3.000 ε, υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το μόνιμο σώμα από 1η Ιανουαρίου 2021 θα πρέπει επίσης ε, να θέσουμε στη διάθεση του μόνιμου σώματος ε, έναν συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων. Το οποίο θα ακολουθήσει τη συνήθη πρακτική, δηλαδή να εντοπιστούν πρώτα οι ανάγκες ε, και λοιπά. Οι ανάγκες, οι δεξιότητες που χρειάζονται και μετά να συνεχίσουμε στην έβρεση του προσωπικού. Θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, δηλαδή EU Agent, δεύτερη κατηγορία ε, National Agents, εθνική υπάλληλοι από τα κράτη-μέλη που θα απασχοληθούν για 2-4 χρόνια και στην κατηγορία 3 θα ανήκει προσωπικό που θα κληθεί να ανταποκριθεί σε περιπτώσεις κρίσης ή έκτακτης ανάγκης. Και τώρα να μιλήσω γαλλικά. Υπήρχε μια ερώτηση για τον τόπο εργασίας των μελών του Ευρωπαϊκού Σώματος. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία 1, δηλαδή τους υπαλλήλους που θα σταλούν από τη Frontex. Ε, προσπαθούμε να εκπονήσουμε τους τρόπους ανάπτυξης των υπαλλήλων αυτών. Θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις όπως κάνουμε σήμερα, το Poseidon, Ποσειδώνας στην Ελλάδα, ε, στην Ιταλία ή στην Ισπανία και άλλες επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις με εκατοντάδες προσωπικό, όπου εκεί μπορούμε να σκεφτούμε ότι για μερικούς μήνες θα σταλεί αυτό το προσωπικό και μετά θα επιστρέφουν στην έδρα για κατάρτιση ε, μερικές εβδομάδες για να πάρουν άδεια για να ξαναδούν την οικογένειά τους ε, και ακολούθω ξαναπηγαίνουν στον τόπο εργασία. Τώρα, για τι μικρότερε επιχειρήσει υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Ε, η ευελιξία είναι η λέξη κλειδί. Ε, ο νομοθέτης, ή μάλλον η Κομισιόν πρότεινε και ο νομοθέτης ενέκρινε αυτή την κατηγορία 1, δηλαδή υπαλλήλων που προσλαμβάνει απευθείας η Frontex, είναι ακριβώς για να έχουμε αυτή την ευελιξία, να χρησιμοποιούμε τα άτομα αυτά εκεί που τα έχουμε ανάγκη. Η επιχειρησιακή, ε, το επιχειρησιακό πλαίσιο θα μας επιτρέπει να, δούμε, να βλέπουμε πού θα έχουμε τις α, ανάγκες. Υπάρχουν εποχιακές ανάγκες, ε, πολύ διαφορετικές από κράτος σε κράτος, ας πούμε. Η ιδέα είναι να στηρίζουμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου Σέγγιν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η μελέτη για τα ευάλωτα σημεία που κάνουμε μας επιτρέπει με βάση και τις μελέτες ε, κινδύνου να δούμε τα είδη των συνόρων, το, το σημείο των συνόρων όπου το Ευρωπαϊκό Σώμα μπορεί να αποσπαστεί και να ε, προσφέρει προσθέμενη αξία για τα τεχνικά στοιχεία. Τώρα, όσον αφορά τον εξοπλισμό μας, σκάφη, αεροσκάφη, τεχνολογικό εξοπλισμό, αυτό ανήκει στην εντολή. Επεξεργαζόμαστε την τεχνολογική στρατηγική για την απόκτηση του εξοπλισμού. Ξεκινήσαμε ήδη με τα οχήματα για τους ε, ελέγχους των συνόρων, των χερσαίων συνόρων. Ετοιμάζουμε πιλωτικό σχέδιο για σκάφη για το 2020. Αναμένεται λοιπόν να ξεκινήσουμε δύο πιλωτικά προγράμματα για να δοκιμάσουμε τέτοια σκάφη ακτοπλοείας και όσον αφορά τις αντιπροσωπείες μας στις διάφορες χώρες θέλουμε να αναθέσουμε τα θέματα επιμελητίας. Έτσι θα αποκεντρώσουμε την διαχείριση των πόρων θα μπορούσε να αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, αλλά θέλουμε και ευελιξία στην τοποθέτηση συνοριοφυλάκων ή επανατοποθέτηση αυτών που μπορεί να είναι καθήκον περιφερειακών αποστολών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι κατάλαβα θα υπάρξει κι άλλη μια συμπληρωματική ερώτηση από την κυρία Στάτλερ, από την κυρία Στρίκ. Σύντομα παρακαλώ, μας τελειώνει ο χρόνος. Μέχρι τις 12, 12 έχουμε πρωινή συνεδρίαση. Και έχουμε ακόμα ένα σημείο στη μέση διάταξη. Είστε σύντομοι παρακαλώ. Με εκπλήσει το ότι ο κ. Τελεζέρ αναφέρθηκε στα θέματα της δίκησης ο αξιωματικός ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι μέλος της διοίκησης, αλλά πρέπει να έχει τεχνογνωσία όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και πρέπει να έχει αυτόνομη θέση. Μπορεί και η διοίκηση να οργανωθεί διαφορετικά. Αν αυτό είναι προτεραιότητα, τεχνογνωσία και ανεξαρτησία όπως είναι στον κανονισμό, συμφωνείτε, δεν εξηγήσατε τη διαδικασία και θα ήθελα Επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί. Και θλίβομαι διότι μετά από ένα έτος θα ξεκινήσει μετά από ένα χρόνο η πρόσληψη ε, εποπτών για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αν είχαμε τον υπεύθυνο θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Ίσως ο κ. Ζέαχ μπορεί να μας εξηγήσει περαιτέρω. Σύντομα παρακαλώ κυρία Στάτλερ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το θέμα την πρώτη εκστρατεία προσλήψεων, 16 Δεκεμβρίου είπατε ότι θα λήξει 3.000 θα απασχοληθούν άμεσα, θα προσληφθούν από την Frontex. Για τον Ιανουάριο, για την κατάρτιση, πόσοι θα συμμετάσχουν. Μετά μία ερώτηση για τον προπολογισμό. Έχετε κάποια αριθμητικά στοιχεία για τον προπολογισμό αν 7.000 άνθρωποι πρέπει να αποσταλούν το κάτι ημέρη, θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα. Πιο μεγάλος προπολογισμό. Έχετε κάποιες ειδήσει όσον αφορά αυτό το θέμα. Κύριε Λεζερή, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, η πρόσληψη των εποπτών δεν θα πρέπει, θα πρέπει να ξεκινήσει στο τέλος του έτους. Θέλουμε να έχουμε στο δυνατόν περισσότερους επιτόπου παρόντες όταν θα αρχίσει η τοποθέτηση του μονίμου συστήματος. Θα αναπτυχθεί από 1η Πρώτου 2021 το μόνιμο σώμα. Όπως εξήγησα, όταν έχεις ένα σώμα, ένα φορέα με 50 ανθρώπους προσωπικό, αυτή είναι η κλίμακα. Είναι λίγο φαϊνότερο διαβάζοντας τον κανονισμό. Λέει 40 επόπτες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ξέρουμε ήδη ότι έχουμε 10 μέλη του προσωπικού στα κεντρικά που ε, ασχολούνται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 50 άνθρωποι λοιπόν. Αν είναι ανεξάρτητος ο φορέα και είναι σαφέστατο αυτό τον κανονισμό ότι υπεύθυνο ο για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανεξάρτητος. Άρα, έχει διοικητικά καθήκοντα. Αλλιώ πώς μπορεί να διαχειριστεί τα 50 μέλη του προσωπικού. Πώς μπορεί να χειριστεί και να προσλάβει τα 50 μέλη του προσωπικού. Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να λυθούν νομικά θέματα, αλλά ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό δεν είναι καθήκον διοικητικό, πέραν από την εξαρτησία και πέρα από τις ικανότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς μπορεί να αμφισβητήσει και να πει ότι δεν είναι διοικητική θέση όταν έχεις πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ προπολογισμό και 50 μέλη που χειρίζεσαι. Εάν συγκρίνουμε με το μέγεθος άλλων φορών του Frontex και, άλλους, και άλλες μικρές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η θέση που συζητούμε δεν είναι διοικητική φύσης. Πρέπει να έχουμε το σύστημα και τον υπεύθυνο αξιωματικό για ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αν ε, δηλωθεί, αν ε, ανακοινωθεί η θέση, θα πρέπει να λάβουμε υποψηφιότητα για να καλυφθεί. Πρέπει να κάνουμε όμως μια διάκριση μεταξύ ατόμων που καλύπτουν θέση και καθηκόντων που εκτελούν σε αυτή τη θέση. Καθήκοντα για τον νομοθέτη είναι σαφέστατο. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ε, είναι ανεξάρτητα τα καθήκοντα, ανεξάρτητη η λειτουργία αυτού του ανθρώπου. Σε αφορά τι προσλήψει, ξέχασα να πω πόσου περιμένουμε για το πρώτο κύμα προσλήψεων. Περιμένουμε να προσλάβουμε από 700 μέχρι 800 για το προσωπικό μας και αναμένεται να υπογράψουν συμβάσεις μέχρι τέλος Μαρτίου ούτως ώστε να ξεκινήσουμε την εκπαίδευσή τους την 1η Απριλίου του 2020 για ένα εξάμεινο. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, αν θυμάμαι σωστά, για του χρόνου περίπου 440 εκατομμύρια ευρώ προτάθηκαν και αναφέρεται στα αναθωρημένα έγγραφα προγραμματισμού που απέστειλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα έστειλα τα έγγραφα και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι βλέπω τα πράγματα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι με την ανάπτυξη του μονίμου σώματος και κυρίως με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που σταδιακά θα αποκτήσουμε να έχουμε και τον κατάλληλο προπολογισμό. Βλέπω αυξανόμενη καμπύλη στον τομέα αυτό Εξαρτάται όμως και από το ρυθμό προσλήψεων. Εάν προσλάβουμε 700 ή 800 αξιωματικούς, δεν θα είναι μεγάλος ο προϋπολογισμός και θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι μεγάλος ο προϋπολογισμός, θα τα καταφέρουμε. Αυτά μπορώ να πω τώρα, διότι θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι και ποιοτικό το προσωπικό που θα προσλάβουμε. Βέβαια, αν προσλάβουμε λιγότερου από του 700-800 θα χρειαστούμε λιγότερα χρήματα. Ευχαριστώ όλου για τις ε, παρεμβάσει σας. Παρακαλώ να μείνετε στην αίθουσα το τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξης πριν αποχαιρετήσουμε τους, το φιλοξενούμενό μας, το Φαμπρί Λεζερή, διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Τώρα, αν αρκεί ο προπολογισμό ή πρέπει να αυξηθεί, αυτό είναι ένα ερώτημα που εν το χρόνο πρέπει να αποφα... αποφασιστεί. Να αποφασιστεί από τις αρχές του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είμαστε εμείς και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριο ε, Οτιάν από τη Renew. Έκθεση για τι κοινωνικέ στατιστικέ για την ε, μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Α ακούσουμε την παρουσίαση τη ε, αναφορά. Πώ θα πάτε με την αναφορά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι συντομότατο. Οι στατιστικέ είναι σημαντικέ για να παίρνουμε σωστέ αποφάσει για την πολιτική και να δίνουμε απαντήσει στι προκλήσει ε, που μα θέτει η μετανάστευση. Γι' αυτό, με μεγάλη χαρά, φτάσαμε σε συμφωνία στον τριμερή διάλογο την περασμένη εβδομάδα και ευχαριστώ του σκιώδει εισηγητέ στην διαπραγματευτική ομάδα για τη στήριξή του. Ε, ο τροποποιημένο κανονισμός επιτρέπει τη συλλογή στατιστικών για τη μετανάστευση υποχρεωτικέ και μιλάμε για 22 νέες δέσμες δεδομένων που έβαλε το Κοινοβούλιο και ψήφισε τελευταία περίοδο. Έγιναν διάφορες ε, συνεδριάσει τριμερού διαλόγου στην Αυστριακή και Ρουμανική Προεδρία με την πρώην ε, εισηγήτρια την κυρία Βίξτρομ που έκανε πολλή δουλειά αλλά δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε πριν τι ευρωπαϊκέ εκλογέ. Η πρώτη ανάγνωση έγινε λοιπόν τον Απρίλιο τελικά και ψηφίσαμε να ξαναρχίσουμε στι 24 Σεπτεμβρίου τι διαπραγματεύσει. και ένα τριμερή διάλογο έγινε ε, στι 28 Νοεμβρίου την περασμένη εβδομάδα και η Φιλανδική Προεδρία μα παρουσίασε κάποιε τεχνικέ αλλαγέ που έγιναν αποδεκτέ από τη ε, διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νέε αναφορικές ε, σκέψεις ε, που δεχτήκαμε. Έγιναν δύο ουσιαστικέ αλλαγέ που συζητήσαμε στον τριμερή διάλογο και συμφωνήσαμε να προσθέσουμε μια νέα αιτιολογική σκέψη και τώρα λοιπόν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την δεύτερη ανάγνωση. Ευχαριστώ για την σύνοψή σας για τις διαπραγματεύσεις για αυτό το θέμα, τις κοινωτικές στατιστικές ε, για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Οι σκιώδεις θα μπορούσαν να πάρουν το λόγο. Δεν βλέπω το σκιώδη της, του ΕΛΚΑ. Ποιος θα τον αντικαταστήσει? Ο κύριος Λέναρτς. Ο κύριος Ορτόλο. Σκιώδης επίσης από τους ε, σοσιαλιστές. Μπορεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος ομάδας μου, ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί ήταν διατεθειμένος να φτάσουμε σε συμφωνία. Ο εισηγητής εξήγησε πολύ σωστά το περιεχόμενο της συμφωνίας που βελτιώνει την κατάσταση σε σχέση με τη σημερινή. Βεβαίω θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα και λάβει περισσότερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε στατιστικές για τις ε, συνθήκες υποδοχής και στατιστικές για τις ε, άδειε παραμονής που ζητούνται για πρώτη χρονιά μέσα τις αντιστοιχές και όχι στις ε, πιλωτικές μελέτες. Παρ' όλα αυτά το συνολικό κείμενο συνολικά είναι καλό, επομένως ε, στηρίζει η ομάδα μου το κείμενο για να κλείσει αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να έχουμε δεδομένα, όχι μόνο επικαιροποιημένα, αλλά τα καλύτερα δυνατά, ούτω ώστε να μπορούμε να νομοθετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κανένα άλλο σημείο. Η κυρία Στρίκ. Και εγώ ήμουν σκιώδη συγγήτρια. Ήρθα σε δύο συνεδριάσεις των σκιωδών ε, εισηγητών. Α, σας ξέχασα βεβαίως και εσείς ήσασταν εισηγήτρια. Συγχαίρω και εγώ τον εισηγητή. Γιατί ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις. Και αυτό το κοινοβούλιο και το προηγούμενο κοινοβούλιο κάνει καλή δουλειά Βάλαμε περισσότερες προϋποθέσεις ό,τι αφορά τα δεδομένα με στον κανονισμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε μόνο με πληροφορίες για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία. Αν θέλουμε να έχουμε μια καλή επισκόπηση για την σωστή εφαρμογή, θα πρέπει να έχουμε δεδομένα τα οποία να είναι συγκρίσιμα και άρα θα πρέπει να έχουμε κριτήρια για αυτά τα δεδομένα, κοινά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα βοηθήσει, το κείμενο αυτό θα βοηθήσει και θα βοηθήσει και το δικό μας ρόλο για να αξιολογούμε το κατά πόσο συμμορφώνονται τα κράτη-μέλη με τους τρέχοντες κανόνες. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτό και σας, σας ε, ελπίζω να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα των πιλωτικών και να τα βάλουμε στον κανονισμό ως ε, διαρθρωτική προϋπόθεση, τα πιλωτικά. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο. Αν όχι, θα ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μας με μια κρόαση σημαντική σήμερα το απόγευμα, από τις 3 και μετά, μέχρι τις 6.30, για μια νέα κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ενίσχυση των εργαλείων και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Από τις 3 και μετά θα γίνει αυτή η ακρόαση.